Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε έστω και με καθυστέρηση. Ε, καθυστερήσαμε λίγο γιατί περιμέναμε τους συναδέλφους που <laughs> δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη. Περιμένουμε τους απόντες. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε κάπως. Πάντως η, η πλειοψηφία είναι εδώ και θα έλεγα να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε τόσο γεμάτο πρόγραμμα. Γι' αυτό και σας ζητώ από τώρα να με συμπαθάτε γιατί θα είμαι πολύ αυστηρό στην τήρηση του χρόνου ομιλίας. Πάμε στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το σημείο 13 του σχεδίου ημερήσιας διάταξης κοινέ διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κτλ. Με αναβάλλεται για τον ε, Ιανουάριο. Ε, κατέτηση της ε, κυρία Ζωανά. Μια και δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Μην ξεχνάτε ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο ε, η συνεδρίαση, 19 γλώσσες διερμηνίας και να εγκρίνουμε βάσει βάση τη διαδικασία ε, τα πρακτικά της 22ης ε, Οκτωβρίου και περνάμε στο κυρίως θέμα, την ε, απαλλαγή για το 2017. Η κυρία Μαριάννα Πετήρ είναι η συντάκτηρα της γνωμοδότησης. Οι συντονιστές είχαμε αποφασίσει να συντάξουμε γνωμοδότηση για την απαλλαγή στο Γενικό Προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, το 2017. Θα δώσω όμως το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Πετήρ, αλλά παρακαλώ χρόνου φίδου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ε, κάθε χρόνο εκφέρει γνώμη για, για το Γενικό Προπολογισμό και την απαλλαγή του. Και αυτή τη φορά ασχοληθήκαμε με τον περσινό προπολογισμό του 2017. Και ω Επιτροπή Γεωργία ενδιαφερόμαστε για την εκτέλεση του προπολογισμού σε ό,τι αφορά τα κονδύλια τη κοινή γεωργική πολιτική. Μεταξύ άλλων, στην γνωμοδότησή μου χαιρετίζω τα απορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου που επιβεβαιώνουν ότι το επίπεδο Σφάλματο εξακολουθεί να μειώνεται από 2,5% το 2016, 2,4% το 2017 στον τομέα φυσική πόρη. Γι' αυτό και ο, ο δημοσιονομικός αντίκτυπος μειώνεται περαιτέρω με δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις, μια και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται στο προϋπολογισμό. Επίσης, η διορθωτική ικανότητα των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων αυξήθηκε στο 2,10% σε σύγκριση με 2,04% το 2016. Επίσης, ε, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι πολύ κοντά και συγκλίνουν με αυτά του ελεκτικού συνεδρίου. Οπότε μπορούμε να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Ε, θα ήθελα να τονίσω δύο ακόμη πράγματα. Καταρχήν, εκφράζουμε τη σοβαρότητα και την ε, επικαιροποίηση των στοιχείων από τα κράτη-μέλη και επίσης είναι σημαντική απλούστευση ε, χάρη στην ε, ηλεκτρονική υποβολή αίτημάτων και υποβολή των στοιχείων. Εμείς θέλουμε να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα, να μειώνονται τα λάθη και τα σφάλματα και επίσης ε, να μην χρειάζεται να δίνουν μάχη με τις διοικητικές διατυπώσεις οι γεωργοί μας και να μπορούν να αφιερωθούν στο έργο τους που είναι η παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων σε προσιτές, τομές, ε, σε τιμές. Και ελπίζω να συμβάλλουμε και στη μεταρρύθμιση του, της ΚΑΠ ε, με τις γνωμοδοτήσεις μας. Αυτή τη φορά ε, μπορούμε να υποβάλουμε και τροπολογίε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση ΚΑΠ στα πλαίσια του νέου πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Γι' αυτό και θα ήθελα να σα παροτρύνω να υποβάλλετε τέτοιε τροπολογίε προς το στο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και να εξασφαλίσουμε μέλλον στη Γεωργία και του γεωργούς μα. Σα ευχαριστώ. Πρώτη, ε, πρώτος γύρος με τους και οδησηγητές, ο κύριος Σάντος, ο πρώτος μας ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι ο σκιώδης εισηγητής, θα μιλήσω εξ ονόματος της συναδέλφου Κάριν Κάντεμπαχ. Οπότε όταν λέω εγώ, εννοώ αυτή εννοεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για το σχέδιο έκθεσης. Είναι καλά τα νέα ότι το Ενεκτικό Συνέδριο ε, επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό λάθους έχει συνεχίσει να μειώνεται και θα είναι ε, κάτω από το όριο ε, της, του ουσιώδους λάθους. Το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε παρόμοια ποσοστά λάθους και στα ε, δύο, και από τα δύο θεσμικά όργανα, παρόλο που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους. Από το ε, Ταμείο Εγγύσεων, ο, ο, το ποσοστό ε, λάθος είναι μικρότερο, είναι 1,92% και το 2017 και το ποσοστό ε, λάθος για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, μια που οι πληρωμές αυτές συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη και εκτείνονται σε ένα φάσμα ετών και περιλαμβάνουν πιο πολλά και πιο περίπλοκα project, το ποσοστό λάθος είναι 3,37%. Παρ' όλα αυτά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης θα πρέπει να βλέπουμε πάντα τι αδυναμίε που προκύπτουν και αν είναι απαραίτητο θα πρέπει να προσαρμοστούν δείκτε ώστε να αποφύγουμε την ε, έλλειψη συμμόρφωση με τι ε, συνθήκε επιλεξιμότητα και να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε καλύτερη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Βεβαίω, προσβλέπουμε στο να αποφεληθούμε από την νέα αυτή προσέγγιση και του νέου δείκτε απόδοση στο μέλλον. Εφόσον βεβαίω θα υπάρξει συνεκτική προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη ώστε να διασφαλιστεί να διασφαλιστούν τα αναμενόμενα από, αυτή την, τομέα πολιτική. Επίση, η, η, η έλεγχη επιτόπου, η καλύτερη, ε, ο καλύτερο έλεγχο των δεδομένων και οι καλύτερε πρακτικέ μπορούν να μα δώσουν καλύτερε πληροφορίε. Σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020 20 πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε στο ποσοστό, το ποσοστό λάθος για να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα ποσοστά λάθος θα συνεχίσουν να μειώνονται και με το νέο πλαίσιο στο μέλλον με αναφορά στις ε, ειδικέ εκθέσεις πάντα στα πλαίσια της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής θα υποβάλω κάποιες σχετικές τροπολογίες. Και επίσης προσβλέπω στην καλή συνεργασία για μια γνωμοδότηση που θα μπορέσει να βοηθήσει να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό λάθος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας θερμά παρακαλώ να είστε λακωνικοί. κυρία Κατάιναν. Ευχαριστώ. Είμαι η σκιώδη συγγήτρια για τους φιλελεύθερους. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την συντάκτρια της γνωμοδότησης για το κείμενό της που είναι πολύ ισορροπημένο και κάνει μια επισκόπηση της Γεωργίας ε, από τη Δημοσιονομική Σκοπιά για το 2017. Χαιρόμαστε που το ποσοστό σφάλματος ε, ακολουθεί τη φθήνουσα πορεία που έχει ξεκινήσει και ελπίζω να μειωθεί περαιτέρω σε ό,τι αφορά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και οι επενδύσει στην αγροτική ανάπτυξη, είναι προγράμματα πολύ θετικά που λειτουργούν καλά και θα πρέπει να συνεχιστούν και να αναδειχθούν στις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, η επιτόπη έλεγχη είναι πολύ σημαντική. Γενικώ είμαστε ικανοποιημένοι με το κείμενο της γνωμοδότησης. Ο κύριος Ντές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Εδώ και πολλά χρόνια ζητώ για το ποσοστό λάθους να γίνουν διαφοροποίησεις για τα λάθη που δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο και για τα λάθη που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει όντω κάποια στιγμή να το διαφοροποιήσουμε, γιατί αλλιώ είμαι πεπισμένο ότι θα είχαμε ακόμη πιο μικρό ποσοστό λάθο. Θα πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουμε ποια είναι τα πραγματικά λάθη και ποια αποτελούν απάτη. Βλέπουμε τι λέει και η έκθεση του ελεκτικού συναδρίου για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα υπάρχουν λάθη που δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Οπότε αυτό θα πρέπει να το δούμε ξεχωριστά. Ευχαριστώ την κυρία Πέτρη για την εξαιρετική της γνωμοδότηση και βεβαίως θα υποβάλω σχετικά και εγώ τη δική μου τροπολογία. Ευχαριστώ. Φυσικά θέλουμε να απλουστεύσουμε τη ζωή των γεωργών. Περί αυτού πρόκειται. κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ την συνάδελφο Πέτυρ για το σχέδιο της γνωμοδότησης. Συμφωνώ μαζί της. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι η εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του ελέγχου αποδίδει καλύτερα και το ελεγκτικό συνέδριο ε, συμφώνησε ότι το 2,4% είναι μια βελτίωση των ποσοστών του σφάλματος. Και επίση ε, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ε, θετικέ προσπάθειε που έχουν γίνει για επίτευξη των ε, στόχων με την ε, πληροφορία, την τεχνική αρρωγή της ε, Κομισιόν προς τις εθνικές αρχές. Θεωρώ πάντως ότι μια απλή καταμέτρηση του ποσοστού σφάλματος δεν συνιστά καθεαυτή αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Και επομένως θεωρώ ότι ακόμα βρισκόμαστε σε υψηλό ποσοστό σφάλματος και έχουμε και τις απάτες μαζί. Άρα κοινοποιήσει ε, και το, το σύστημα προς τα κράτη-μέλη, το σύστημα των κοινοποιήσεων φύγεται από τα λάθη. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο στη συνέχεια. Ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο κ. Μέγκελε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, την Επιτροπή Άγκρη, για τη γνωμοδότηση που συνέταξε. Το έργο επί της γνωμοδοτήσεως έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και είναι σημαντικό ε, να ακούγεται η φωνή του γεωργικού κόσμου στη συζήτηση για την απαλλαγή. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Χαιρετίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης κυρίας Πετήρ. Η συγγήτρια πολύ εύστοχα παρουσίασε τα εξαιρετικά αποτελέσματα που υλοποίησαμε κατά το 2017. 2,4% είναι το γενικό ποσοστό σφάλματος ε, που επισημαίνει και το ελεκτικό συνέδριο και θα ήθελα να τονίσω ότι ο πρώτος πυλώνας που είναι το κύριο τμήμα των πληρωμών ε, είναι κάτω από 2% το ποσοστό σφάλματος. Εκεί είναι που γίνονται οι περισσότερες πληρωμές, εκεί είναι τα περισσότερα κονδύλια και εκεί είναι... είμαστε πράσινοι, όχι πράσινοι λόγω της γεωργίας, αλλά γιατί έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Επίσης θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι αυτό δεν είναι ε, κάτι ουρανοκατέβατο, ούτε κάποιο θαύμα. Προέρχεται από τις προσπάθειες των κρατών μελών και την ε, ε, επιδείξει Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τη διαχείριση και τους ελέγχους. Η πιο αυστηρή έλεγχη και οι αυστηρότεροι κανόνες οδηγούν βέβαια σε αυξημένο διοικητικό φόρτο. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε κάποιες προτάσεις μεταρρυθμίσεων που στόχο έχουν να διαρρήξουν αυτό το φαύλο κύκλο των όλο και αυστηρότερων κανόνων και ελέγχων και όλο και περισσότερου δι διοικητικού άχθους. Προσπαθούμε λοιπόν να μεταφέρουμε την έφαση από την κανονικότητα και την νομιμότητα στις επιδόσεις, στα αποτελέσματα δηλαδή. Μεταστρέφουμε το ενδιαφέρον μας προς τα αποτελέσματα που θέλουμε από την ΚΑΠ και όχι τόσο την νομιμότητα και την κανονικότητα. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αργότερα όταν θα συζητηθεί ο οριζόντιος κανονισμός και η σχετική έκθεση. Ευχαριστώ και πάλι θερμά την Επιτροπή σα για την γνωμοδότησή τη που θα μα βοηθήσει πολύ στη γενική διαδικασία τη απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φλάναγκαν ζήτησε το λόγο. Δεν είχατε δηλώσει εγκαίρω το ενδιαφέρον σας να μιλήσετε, γι' αυτό και έδωσα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά έχετε το λόγο κύριε Φλάναγκαν. Είναι αρκετά σαφής αυτή η ερώτηση για το όσα είπε ο κύριος Μέγκελε. Νομίζω ότι πρέπει έτσι θερμό να απαντήσουμε. Ε, ίσως έτσι να πρέπει να δουλεύει η Επιτροπή. Συγγνώμη, εν πάση περιπτώσει, αν το κάνω. Αλλά αν τα συστήματα που βελτιώνονται συνέχεια και λειτουργούν όλο καλύτερα, γιατί να τα αλλάξουμε. Μιλάτε για το διοικητικό άχθος τον, το ογκώδες διοικητικό άγχος. Από την νέα πρόταση της ε, γεωργική πολιτική φαίνεται ότι το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι το διοικητικό άγχο θα φύγει από εδώ και θα πάει στο Δουβλίνο και γενικώ στις πρωτεύουσε όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Οπότε, τι ακριβώς κάνουμε εδώ. Μια μετακύληση του άχθους. Πώς θα μπορέσετε εσεί να μετρήσετε με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο που το κάνουμε τώρα, αν φύγει από εδώ το άχθος, από το κέντρο και πάει στις πρωτεύουσες των κρατών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέγκελε παρακαλώ αν μπορεί να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική που ε, κάθε χρόνια ε, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται 80 δισεκατομμύρια, ε, δεν μπορεί να μην έχει διοικητικό άκθο. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε να το μειώσουμε αυτό το άκθο. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική, αυτό που προσπαθεί να επιτύχει είναι να μειώσει τι λεπτομέρειε στου κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι σύντομες, περιληπτικοί οι κανόνες, ε, να ε, περιορίσουμε ας πούμε τον αριθμό των δέντρων που επιτρέπονται, πόσο ε, πλατής πρέπει να είναι οι φράχτες κλπ. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε λίγο πιο κοντά στο τι συμβαίνει πραγματικά επιτόπου. Και θέλουμε να έχουμε κανόνες που όντως θα ταιριάζουν και στα νομικά συστήματα και τα διοικητικά συστήματα των κρατών μελών και θα είναι και πιο στοχευμένοι για να πετύχουν τελικά τα αποτελέσματα που θέλουμε. Άρα λιγότερους ελέγχους στα, α, στις επιτόπου α, περιοχές. Το θέμα είναι αν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε. Όχι να συζητούμε κάθε μέρα, κάθε φορά αν όντω έχει εφαρμοστεί, αν έχει μεταφερθεί σωστά κάθε μικρή λεπτομεριούλα. Σας ευχαριστώ. Η συγγετριά μας τώρα, η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά της. Θα έλεγα ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι προχωράμε. Και ε, ήδη περιμένω με χαρά και ανυπομονησία τις τροπολογίες που πιστεύω θα βελτιώσουν τη γνωμοδότηση που οι συνάδελφοι ήδη έκριναν θετικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την συντάκτρια. Ε, μέχρι τις 27 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι μπορείτε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας. 27 Νοεμβρίου, μία το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Και πάμε στο επόμενο σημείο, το 5 χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Όπως ξέρουμε, η συγγήτρια είναι η κυρία Μίλλερ. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τους καλεσμένους κυρίες Μίλλερ. Γεωργούς από, το γεωργικό, από ένα γεωργικό συνεταιρισμό της Βαβαρίας. Καλώς ήρθατε. Θα ακούσετε μια πολύ σημαντική συζήτηση που θα κάνουμε για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μίλλορ για να μας παρουσιάσει πρώτα την έκθεσή της και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ας περάσουμε κατευθείαν στην παρουσίαση της έκθεσης. Κυρία Μίλλερ, έχετε το λόγο. Τα διαφανή θεσμικά όργανα και οι απλουστεύσεις ε, είναι τα βασικά σημεία που έχω στην πρότασή μου για αυτόν τον οριζόντιο κανονισμό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Αγαπητέ κυρίες και κύριοι. Ε, χαίρομαι που μπορώ σήμερα να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου για την ε, διαχείριση, χρηματοδότηση και εποπτεία της κοινή γεωργική πολιτική οριζόντια, όπως λέει το όνομα, οριζόντιος είναι ο κανονισμός αυτός και βεβαίως έχει άπτεται και των τριών αυτών θεμάτων, κυρίως όταν μιλούμε για την εκπόνηση των νέων στρατηγικών σχεδίων, τις άμεσες πληρωμές δηλαδή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ο οριζόντιος αυτός κανονισμός βασίζεται φυσικά στις, στους δημοσιονομικούς κανονισμούς που αποτελούν βεβαίως τη βάση όλων των προγραμμάτων δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος μου είναι για τη Γεωργία να έχουμε ένα νομικό κείμενο το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια για τους κανόνες ε, ε, εφαρμογής και θα αποτελεί απλούστευση στην εφαρμογή τους. Γι' αυτό, μετά τι πρώτες συζητήσει τον Ιούλιο στην Επιτροπή Γεωργίας, συναντήθηκα με τους προσώπους της Κομισιόν, με τους ε, σκιώδει ηγητέ και με τους εισηγητέ των τεσσάρων επιτροπών που θα κάνουν γνωμοδότηση και συναντηθήκαμε μάλιστα τέσσερι φορέ. Επίση. Ε, ζήτησα μία μελέτη από την Οικονομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου για να δούμε λιγάκι τις ε, διοικητικέ δομές των κρατών μελών. Δυστυχώ, δεν κατάφερα με την, ομάδα, με την ε, μελέτη αυτή να καλύψω όλα τα κράτη-μέλη και τα 28. Διαλέξαμε τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, επειδή έχουν περιφερειακά προγράμματα, την Ιρλανδία, τι κάτω και τη Ρουμανία. Τα αποτελέσματα αυτή τη μελέτη. Ε, τα ανακοίνωσα στην τελευταία συνάντηση στους, τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο στους και οδησηγητές. Επίσης άλλο ένα, άλλη μια εξωτερική έκθεση ήταν η εκνομοδότηση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Χαίρομαι πολύ για την ανταλλαγή απόψεων που θα κάνουμε και τη συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Και τώρα θα σας πω λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την έκθεσή μου Έχω 7 σημεία συγκεκριμένα που θέλω να σας παρουσιάσω. Καταρχάς, το κεφάλαιο 2 για την ε, απλούστευση των ε, διοικητικών δομών. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί το, ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας θα συγχωνευτούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις συνέργειες που υπάρχουν και να ξεκαθαρίσουμε τις επικαλύψεις. Γι' αυτό, για παράδειγμα, για τις διοικητικές αρχές, άρθρο 110 των στρατηγικών σχεδίων και την Συνοδευτική Επιτροπή, άρθρο 111, θεωρώ ότι πρέπει να, μπει, να μπουν πίσω στον ε, ε, γενικό κανονισμό για να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματικέ διοικητικέ δομέ για τα κράτη-μέλη. Για τι άμεσε πληρωμέ θα πρέπει στο μέλλον να υπάρξει και άλλη μια ε, επιτροπή παρακολούθηση η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για την αναπτύξη τη υπαίθρου. Νέοι τομεί τώρα. Για την πιστοποίηση υπάρχουν και τι πιστοποιητικέ αρχέ στα, στο νέο σύστημα θα έχουν πολύ περισσότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ως προς αυτό παραπέμπω στο προηγούμενο άρθρο 7 για τις άλλες δαπάνε συμπεριλαμβανομένων και, τη τεχνική βοήθεια. τεχνικής στο σχέδιο ε, ΚΚΠ 111. Ε, από τα υπάρχοντα μέλη λοιπόν, ε, ε, κονδύλια συγγνώμη, μιλάμε για ένα πιο υψηλό ε, ποσοστό για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα κονδύλια και να εγγυηθούμε καλύτερη εφαρμογή. Επιπλέον, ο στόχο μου ήταν με τι τροπολογίε μου στον κανονισμό αυτό τα συγκεκριμένα, τις συγκεκριμένες ομοσπονδιακές δομές των κρατών μελών να τις λάβουμε επαρκώς υπόψη. Το θέμα της επικουρικότητας επίσης είναι σημαντικό για όλους και στο κεφάλαιο 2 είναι πραγματικά τόσο περίπλοκος το τομέας αυτός που θα ήθελα και οι συνάδελφοι να το διαβάσουν πολύ προσεκτικά Γι' αυτό και για να μπορέσουν να καταλάβουν τι ιδέε και τι τροπολογίε μου. Σημείο 2. Ε, οι συμβουλευτικέ υπηρεσίε για, την, ε, τη γεωργία. Θεωρώ ότι είναι μια καινοτομία αυτή για την βιωσιμότητα τη δασοπονία και τη γεωργία για το μέλλον. Για το λόγο αυτό, ανήκει στον οριζόντιο κανονισμό και αυτό το σημείο και θα πρέπει να αναπτυχθεί με περισσότερες λεπτομέρειες και να ληφθεί υπόψη στις ε, διαθεσμικές ε, υπηρεσίες. Η υπηρεσία αυτή επίσης ε, θα περιλαμβάνει και την ανταλλαγή πληροφοριών γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Τώρα, το πώς οι γεωργοί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν πρόσβαση στα καλύτερα συστήματα και σε συμβουλή για τη γεωργία αλλά και για θέματα έρευνας. Επίση, τα αποθεματικά για τι κρίσει. Σε περιπτώσει όπου οι πιθανότητε για ύπαρξη κρίση είναι πολύ ψηλέ, θα πρέπει να έχουμε ένα καλό λειτουργών και ανεξάρτητο σύστημα διαχείριση κρίσεων και γι' αυτό προτείνω ένα αποθεματικό για τις κρίσεις, αποκλειστικά για τη χρήση σε περίπτωση κρίσης και όχι για παρεμβάσεις στην αγορά. Επίσης, να θυμίσω τι, έγινε την, στην τελευταία φορά που είχαμε κρίση. Είδαμε ότι τα χρήματα δεν έφταναν και όταν ε, θέλαμε να πάρουμε τα λεφτά από τους ε, γεωργούς και να τα ξαναδώσουμε για να καλύψουμε τα έξοδα της κρίσης ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο γιατί σίγουρα ε, είναι σαν να τιμωρούμε τους γεωργούς δύο φορές. Τρίτον, οι, τα υποχρεώσει υποβολή εκθέσεων. Στι τροπολογίε μου, στην 150 συγκεκριμένα για το άρθρο 52 τη Κομισιόν, η πρόταση της Κομισιόν λέει ετήσια έκθεση ε, η μου, το δικό μου το σκεπτικό είναι αυτή η ετήσια υποχρέωση να γίνει διετής, να αλλάξει η υποχρέωση αυτή. Ελπίζω η, η Γκαρσία να συμφωνεί με αυτό. Να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που δεν θα επικεντρώνεται μόνο στο output, αλλά ε, αλλά θα, ε, θα βασίζεται και στο output και στα αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί να είναι θετικό. Και επίσης θεωρώ ότι το, οδηγητικό άχθος αυξάνεται συνεχώς και η σκοπιμότητα αλλά και η ποιότητα των ε, νέων αυτών, του νέου αυτού συστήματος θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε μόνο αν κάνουμε προσαρμογή αυτού του κύκλου εκθέσεων από ένα έτος σε δύο έτη. Δυστυχώ όταν ε, υποβάλαμε το κείμενο έχει, έγινε και ένα ε, ε λάθος τυπογραφικό. Λέει το κείμενο κάθε εξάμεινο. Όχι, θα διορθωθεί το λάθος αυτό και θα λέει δύο έτη. Κάθε δύο έτη έκθεση απόδοσης. Πέμπτο σημείο είναι ο καθορισμός των κυρώσεων. Στο άρθρο 85 και 86 ως περαιτέρω απλούστευση προτείνω το κατόφλι για τις εξαιρέσεις για τις κυρώσεις από 250 ε, ευρώ ε, και για 10 εκτάρια γιατί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διοίκηση και για, από την πλευρά των Γεωργών. Επίσης, ε, μπορούν να, μπορεί να ενισχυθούν οι επιτόπου έλεγχοι και να ληφθούν υπόψη από τα κράτη-μέλη. Επίση, τα δεδομένα που έχουμε από του δορυφόρου μπορούν να βελτιωθούν και να οδηγήσουν σε καλύτερου ελέγχου. Και επίση, για να έχουμε πιο πολύ ομοιογένεια, θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό σύστημα για την βαθμιδόν επιβολή κυρώσεων. Βεβαίω, θα πρέπει να δούμε και τι παραβάσει. Εγώ προτείνω να υπάρξουν ποσοστά. Ως προς αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η διατήρηση της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρέπει να έχουμε ε, χαμηλότερα ε, ποσοστά σε σχέση με τον τρέχοντα κανονισμό. Έκτο σημείο είναι ε, οι εκτελεστικέ πράξεις και η κατεξουδότηση πράξεις. Στον οριζόντιο κανονισμό υπάρχουν συνολικά 100 εκχωρήσει προς την Κομισιόν για 104 άρθρα. Μιλούμε για 70 πράξεις εκτελεστικές και 30 κατεξιοδότηση. Για την έκθεση αυτή μελετήσαμε μια έκθεση από το 2013 για τα κριτήρια διαχωρισμού για τις ε, κατεξουδότηση και α, α, εκτελεστικές πράξεις. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή αυτή, αυτή αυτές οι 35 τροπολογίες υπευλήθησαν. Η Κομισιόν λέει ότι συνολικά 50% λιγότερες ε, κατεξουδότηση και εκτελεστικές πράξεις θα έχουμε πλέον στον οριζόντο κανονισμό. Όμως αυτό δεν φαίνεται. Επίσης ε, θα ήθελα περισσότερο, ε, να ρυθμίζονται περισσότερα πράγματα στο διατακτικό του κειμένου, του κανονισμού, αλλά ως προς αυτό δεν έχουμε αρμοδιότητα και δεν υπάρχουν και οι πόροι ώστε εδώ να μπορέσουμε να ε, συγγράψουμε τον, το, τον όγκο του κανονισμού. Και επίσης οι μεταβατικές περίοδοι οι προθεσμίε για την ε, θέση ε, εφαρμογή των νομοθετικών ε, πράξεων θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο τελευταίο, στην τελευταία προγραμματική περίοδο είχαμε διετή μεταβατική περίοδο. Αυτό λείπει γιατί πλέον δεν καλύπτει ούτε την λήξη της θητείας της Κομισιόν ούτε την έναρξη νέων δομών. Οπότε, τίθεται το ερώτημα τι κάνουμε, φτάνει το νησιν 2, μήπως χρειαζόμαστε νησιν 3 ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, το Omnibus και τις δυνατότητες από εκεί ε, και να συνεχίσουμε μέχρι να έχουμε μια νέα συνολική κοινή γεωργική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει έγκυρα να αντιδράσουμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια βεβαιότητα για τα κρατη και για τους γεωργούς. Κλείνοντας, να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι για ε, για εμάς θα πρέπει να υπάρξει όσο δυνατόν περισσότερη ε, απλούστευση για τις ε, διοικητικές δομές αλλά και για την λήψη αποφάσεων. Χαίρομαι λοιπόν για την ε, ανταλλαγή απόψεων και με εσά και με την Κομισιόν και βεβαίως θα δούμε από κοινού τις τροπολογίες που θα υποβάλλετε. Ευχαριστώ. Όπως είπαμε θα ακούσουμε πρώτα τους και ηγητές και θα σας ήμουν ευγνώμων αν καταφέρετε να ολοκληρώσετε μέσα σε ένα λεπτό τα σχόλιά σας. Ο κύριος Νταντά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της, για τη συνεργασία μας όσον αφορά το κείμενο και είναι σημαντικό που σήμερα η ΚΑΠ δικαιώνεται και υπάρχουν εγγύσει, ισότητα μεταχείριση για τους ε, γεωργού σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτέ είναι οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι γεωργικέ εκμεταλλεύσεις. Μα γι' αυτό και εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω από τα όσα προτείνει η συγγήτρια. Να έχουμε κάποιου άλλου κοινού κανόνε για τους ελέγχους, τις χρηματικές ποινές, την ανάκτηση των ε, οφειλωμένων. Οπότε, λάβουμε υπόψη τα όσα για τους τελευταίους μήνες, θα πρέπει να οριστεί ποια, ποια είναι τα γεγονότα που συνιστούν ε, ανωτέρα βία. Μα δεν είναι κλέφτες οι γεωργοί. Είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι, ότι ωφελούνται από τα λάθη, κερδίζουν, κερδίζουν από αυτά και γι' αυτό και θα πρέπει να τους σταυρώσουμε. Ούτε είναι δυνατόν να επιβαρύνονται υπερβολικά από ελέγχους. Γιατί βλέπουμε επανειλημμένα ότι τα περάσματα για τις αγελάδες είναι πάρα πολύ στενά σε κάποιο λιβάδι. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να επιβαρυνθούν. Ε, θα πρέπει τέτοιοι κανονισμοί να διορθωθούν. Δεν θα πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε την ε, ρύθμιση και λάβαμε υπόψη το, ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να είναι το σύστημα πιο κατανοητό και ε, αυτό θα δει σε καλύτερες επιδόσεις. Λέει για έκθεση αναδιατία εισηγήτρια που να λάβουμε υπόψη τι είπε η συνάδελφος Καρτία για τον πρώτο πυλώνα. Έχουμε το στρατηγικό πρόγραμμα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα πλαίσια αυτού τα όσα ισχύουν στον οριζόντιο κανονισμό για τους ελέγχους. Άρα αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε, το στρατηγικό πρόγραμμα, για να δούμε τι θα κάνουμε με τον οριζόντιο κανονισμό. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μίλλερ για το διαφανή τρόπο και το πολύ επικοδομητικό πνεύμα που χαρακτήρισε τις συναντήσεις με τους κοιόδης ηγητές. Η πρόταση αυτή διατηρεί πολλές διατάξεις του τρέχοντος κανονισμού ε, και παρόλα αυτά περιλαμβάνει κάποια καινοτόμα στοιχεία σε ό,τι αφορά το νέο μοντέλο, το delivery model παροχής αποτελεσμάτων δηλαδή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το νέο delivery model ε, θα αυξήσει κατά τη γνώμη μου το διοικητικό φόρτο των εθνικών διοικήσεων και αναγκαστικά θα επιρρηθεί αυτή η αύξηση του διοικητικού άκθους και στους ε, αγρότες. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα της πρότασης. Κυρίως ε, η διασύνδεσή της με την πρόταση κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια, γιατί είναι αλληλεύθετα τα δύο θέματα. Για παράδειγμα, έχουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης. Ε, η δομή, ο σκελετός αυτού του συστήματος έχει διαφυλαχθεί. Ε, και η προσαρμογή του στο νέο μοντέλο δεν προσδιορίζεται σαφώς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των διαφόρων φορέων, φορέων πληρωμής, ε, φορέων συντονισμού, αρμόδιων αρχών, γιατί αυτό περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια ποιος είναι ο ρόλος τους και πώς ε, συνεργάζονται ή διαρθρώνονται οι διάφορες αρχές και οι διάφοροι φορείς σε ό,τι αφορά την, ε, την υποβολή των εκθέσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ασφάλεια δικαίου για να μην υπάρχουν ασάφειες ούτε για τις διοικήσεις ούτε για τους γεωργούς. Επίσης, ναι, αναφέρεται το θέμα της χρηματοδότησης του γεωργικού αποθεματικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συσταθεί το αποθεματικό από τα κονδύλια που περισσεύουν από τον κάθε ετήσιο προϋπολογισμό. Ε, βέβαια την περισμένη εβδομάδα ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε 450 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, για την σύσταση του αποθεματικού που είναι επιπλέον ποσό σε σχέση με τον ε, γεωργικό προϋπολογισμό της ΚΑΠ για την επόμενη, ε, την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Έτσι θα διαφυλάξουμε τα κονδύλια της ΚΑΠ και θα επιστρέψουμε τα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους που είναι οι γεωργοί. Αυτά προς το παρόν και ελπίζω να συνεχίσουμε την καρποφόρα συνεργασία με την εισηγήτρια και του και εισηγητές, ώστε αυτόν τον αμυγό ιδιαίτερα τεχνικό προπολογισμό να το φέρουμε σε αίσιο, το κανονισμό, συγγνώμη, να το φέρουμε σε αίσιο πέρας. Χόιμπουχ. Όπως ξέρετε, ίσω, εγώ είμαι από την... Θα προσπαθήσω μάλλον να συνοψίσω λίγο τις ε, τα σχόλια και από την Επιτροπή ανάπτυξη. Ε, εγώ ε, ήμουνα σε, έναν κοινό, σε μια κοινή συνάντηση με του εμπειρογνώμονε. και επίσης πρόσεξα τι έκανε η Επιτροπή Ανάπτυξης για τον κανονισμό αυτό από το 2011, γιατί και τότε υπήρχε μια έκθεση, μια γνωμοδότηση της Επιτροπής ανάπτυξη από μια συνάδελφο από το ΕΛΚ και η γνωμοδότηση αυτή τη συναδέλφου τη Γερμανίδα από το, από το Τσεντεού ε, ξεκίναγε από την οπτική τη ε, αναπτυξιακή πολιτική. Θα πρέπει να έχουμε μια τελείω διαφορετική ε, γεωργική πολιτική σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει ειλικρινώ να πω ότι αυτή την ε, φράση, με αυτή τη φράση συμφωνώ απόλυτα γιατί η κοινή γεωργική μας πολιτική έχει πραγματικά πολύ, σημαντικές, ε, ε, πολύ σημαντικό αντίκτυπο κυρίως αν σκεφτούμε τι εξαγωγέ προ την Αφρική, για τα πουλερικά, αν δούμε την βιομηχανία στην Ευρώπη, αν δούμε τι γίνεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τι γίνεται με τους γεωργούς στις αναπτυσσόμενες χώρες που υποφέρουν από όλε αυτές τις αλλαγές και βεβαίω οι κυβερνήσεις τους ελάχιστα ε, μέσα έχουν για να τους ε, προστατεύσουν. Και μπορεί να μην έχουν καν και το ενδιαφέρον να το κάνουν. Οπότε ε, θα κάνω κάποιες προτάσεις για τον οριζόντιο κανονισμό. Καταρχάς, θέλω μια, ένα συστηματικό έλεγχο, μια υποπτία των, ε, του αντικτύπου της ε, ε, γεωργικής πολιτικής στην ε, ανάπτυξη. Γιατί προς το, προς το παρόν, παρόλο που έχουμε από μεθοδική πλευρά τη δυνατότητα να το, να το πράξουμε, δεν έχουμε ουσιαστικά δεδομένα. Έχουμε ε, στοιχεία από τις χώρες εταίρους και θέλουμε να τα ζητούμε. Είναι σημαντικό όμως να δούμε τι οικονομικό, οικονομικό αντίκτυπο στα κράτη-μέλη όταν δεν σέβονται την αρχή αυτή για το πώς δηλαδή μπορούν να συνδυαστούν η γεωργική πολιτική με την αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί μιλούμε για συνοχή των πολιτικών που πρέπει πάντα να τηρείται και επίσης ε, είμαι αρκετά διστατική για αυτή την μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής ε, γιατί πρέπει να την ε, καταστήσουμε φιλική προς τους χρήστε. Την τελευταία φορά είδαμε ότι έγιναν πολλά μέσω των μεταρρυθμίσεων, είχαμε μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015 και δόθηκε πολύ μεγάλη προσοχή στα θέματα αναπτυξιακή πολιτική. και στην έλλειψη συνοχής των πολιτικών. Από τότε βέβαια η έλλειψη αυτή έχει αυξηθεί. Ο Επιτρόπος Χόγκαν έχει μια task force για την Αφρική ε, έχει δημιουργήσει μια task force η οποία δουλεύει πάνω σε συστάσεις και για αυτή τη μεταρρύθμιση και έχουμε μία παράγραφο, την 208 της Συνθήκης Λισαβόνας και την υποχρέωση από εκεί να είμαστε συνεκτικοί στις πολιτικές μας με τις, αναπτυξιακές, με τις χώρες. Οπότε παρακαλώ αυτή την κοινή, αυτή τη μεταρρύθμιση ας την καταστήσουμε λίγο πιο φιλική και για τα θέματα αναπτυξιακής πολιτικής. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο μιλίας που δικαιούστε. Ο κύριος Μάρκο Τζούλο, παρακαλώ. E Ευχαριστούμε την εισηγήτρια σε συντομία. Ολοκλήρωσε αυτή την έκθεση εντελεχώ. Οπότε η μεταρρύθμιση της διακυβέρνηση για την ε, ΕΚΑΠ είναι απαραίτητη για να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία, κυρίω με αυτή την καινούργια φιλοσοφία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι σχετικά με τις ε, επιδόσεις, αλλά τώρα είναι πιο στεγανή η αρχιτεκτονική και έχουν πιο αποτελεσματικούς ελέγχους, οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ποιες είναι οι προβλεπόμενες ε, αλλαγές. Και στην Ιταλία και σε άλλες ε, χώρες τώρα έχει αποδειχθεί ότι δεν αποδίδουν οι έλεγχοι, ότι υπάρχουν κενά και πολλές φορές έχουμε φαινόμενα παρανομίας. Αυτό είναι δυσλειτουργία και αυτό είναι κακό για την δημοσιονομική πειθαρχία στην ΚΑΠ και έχουμε καθυστερήσεις, εμπόδια για τους γεωργούς, οπότε δεν υπάρχει σιγουριά στα αυτά που πρέπει να εισπράξουν. Από θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αρμοδιότητες της Κομισιόν και των κρατών μελών, ε, να δούμε τώρα αυτό το καινούργιο delivery model τι θα προβλέπει και θα πρέπει να δούμε πως υπάρχουν βελτίωση, υπάρχει βελτίωση τώρα στα πράγματα. Οπότε αυτοί οι νέοι θεσπιζόμενοι κανόνες θα, πρέπει να δούμε αν βγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση, την αποτελεσματικότητα. Ε, τέλος πάντων, ό,τι στρεβλώσεις υπάρχουν θα πρέπει να φέρουν κάποια διόρθωση πορείας. Ο κύριο ε, Φιλίπ Λουαζό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Μίλλερ, την εισηγήτρια. Στο κείμενο ε, γίνεται λόγος για μια έξυπνη γεωργία. η ε, Ευρωπαϊκή Γεωργοί και κυρίως οι Γάλλοι Γεωργοί θα ήθελαν και μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν θα είναι αντιφατική, που δεν θα απαιτεί υπερβολικές ε, περιβαλλοντικές διατάξεις ε, και θα τους επιβάλλει στους γεωργούς και φυσικά θα δίνει έμφαση σε, στην ε, τοπική αλυσίδα παραγωγής και δεν θα ευνοεί τα εισαγόμενα προϊόντα που έρχονται από μεγάλες αποστάσεις. Και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να προσπαθεί να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και αυτό που χαρακτηρίζει πρόοδος, τι να σας πω, λέει να εξασφαλίσει ε, δίκαιο βιωτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό με την ε, αναβάθμιση του ατομικού εισοδήματο. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη ε, τα, τις ΜΕΤ, τα, ανησυχίες των Γεωργών, τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, τα προβλήματα στο γαλακτοκομικό τομέα, τις κρίσεις που πολλαπλασιάζονται και τίποτα δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τους Γεωργούς. Στο άρθρο 39, ένας από τους στόχους ε, της ΚΑΠ ε, είναι η εξασφάλιση δίκαιου ε, η κατάλληλου βιωτικού επίπεδου στους γεωργούς. Με ποιο τρόπο σκοπεύει να το υλοποιήσει αυτό το στόχο της ΚΑΠ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε στους υπόλοιπους συναδέλφους, μια και έγινε ένας γύρος με τους σκιώδεις ηγητές. Μην ξεχνάτε ότι στη συνέχεια θα εξετάσουμε την έκθεση τη κυρίας Εράς Γκαρσία για τα στρατηγικά σχέδια δηλαδή. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να επεκταθείτε και στη δεύτερη συζήτηση. Ένα λεπτό καθένα, Ο κύριος Αρντός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία εισηγήτρια, τρεις ε, παρατηρήσεις έχω για την έκθεση. Καταρχά, οι εκχωρήσει ε, αρμοδιοτήτων προς την Κομισιόν θα πρέπει να περιοριστούν σε ό,τι αφορά την, θα πρέπει να αποφύγουμε υποκειμενικές αποφάσεις. Δεύτερον, υποστηρίζω την διετή αυτή υποβολή εκθέσεων, αλλά παραμένει ένα ερώτημα με αυτή θα γίνεται και εποπτεία κάθε δύο χρόνια και θα υποβάλλεται η έκθεση κάθε δύο χρόνια. Αυτή είναι η πρότασή μου. Και τρίτον, για την ανάπτυξη πέθρου, το νη συν 3 ε, θα ήθελα να διατηρηθεί. Γιατί με τα προγράμματα των επιδοτήσεων μπορεί να υπάρξουν και κάποια έκτακτα γεγονότα. Οπότε χρειαζόμαστε να έχουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπράβο σα. Ιδανική η διάρκεια του χρόνου ομιλία σα. Η κυρία Ρα Γκαρσία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μίλλερ για το έργο τη. Από αυτό που μα είπε σήμερα, αυτό που με προβληματίζει ή που μου τραβάει την προσοχή είναι ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε την εφαρμογή του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια. Δεν φαίνεται όμως ότι τη διευκολύνουμε ε, την εφαρμογή του κανονισμού στρατηγικών σχεδίων αν περάσουμε στον οριζόντιο κανονισμό το θέμα ε, των αρμόδιων διχειριστικών παραγόντων της Επιτροπής Παρακολούθησης και των άλλων συμβουλευτικών επιτροπών. Νομίζω ότι περισσότερο έχουν θέση στον κανονισμό στρατηγικών σχεδίων. Σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις επιδόσεων, ξέρω ότι και ο κύριος Νταντά είναι υπέρ του πολιετούς χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα διοικητικό ζήτημα. Αυτό που θέλω είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και να μην ε, τα τιμωρήσουμε και να μπορούν να αντιδρούν εγκαίρως. Αν θεωρείτε το πολιτέ σύστημα είναι καλύτερο να το συζητήσουμε. Πάντως θα ήθελα να πω ότι θα καταθέσω μια τροπολογία για το αποθεματικό κρίσεων, ώστε τα ε, κονδύλια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί να μένουν για την επόμενη χρονιά, ώστε να μην πλήξουμε τους γεωργούς και να μην ε, στερήσουμε από τις επόμενες χρονιές τα δικαιώματα των γεωργών. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ την συνάδελφο Μίλλερ για την εξαιρετική δουλειά της, είναι δύσκολη για, λόγω όλων αυτών των χαρακτηριστικών της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε σχέση με τις αρμοδιότητες αυτής και των κρατών μελών πρέπει να δούμε τι πρέπει να προσεχθεί εδώ πέρα. Πρώτα πρώτα οι οργανισμοί, οι καταβάλλοντες, οι οργανισμοί που ασκούν την ε, διαχείριση χρειάζεται μεταξύ αυτών των συναρμοδίων οργανισμών να υπάρχει περισσότερο συντονισμό σε κάθε περιφέρεια και επίσης για τα στρατηγικά σχέδια να υπάρχει οργανισμός διαχείρισης Οπότε θα πρέπει μέσα στην κρίση να υπάρχει κάποια αρρωγή ή υποστήριξη. Άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε τους ε, μηχανισμούς ε, κρίσης που να έχουν σε αυτήν την κρίση ως μοναδική αρμοδιότητα και όχι άλλες παρεμβάσεις. Επίσης, πρέπει να δούμε τι γίνεται με κυρώσεις και ελέγχους και να δούμε τα σχετικά ποσά. Ε, βλέπω είναι αρκετά χαμηλά. Και επίσης θα πρέπει να δούμε αυτό το κριτήριο της επιφανείας του εμβαδού για αυτές τις κυρώσεις. Και πρέπει τα κράτη μέλη να πάρουν τα δορυφορικά δεδομένα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλούμε για την ΚΑ Πρόεδρε. Συμπάθαμε, αλλά μιλάμε για τη μεταρρύθμιση αυτής. Και είναι το μοναδικό θέμα για το οποίο έχουμε εδώ αρμοδιότητα. Ε, αλλά ε, μας περιορίζεται πάρα πολύ. Ε, άμα είναι έτσι, το ανησυχωθούμε να φύγουμε. Δεν, δεν μπορούμε να συζητήσουμε στην ΚΑΠ, δεν μπορούμε να συζητήσουμε στην, στην Επιτροπή, δεν μπορούμε να συζητήσουμε στην Ολομέλεια. Ε, πότε θα συζητήσουμε. Δύο λεπτά μιλήσατε. Είπαμε ένα λεπτό. Κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μίλλερ για την έκθεσή της. Σίγουρα μερικές προτάσεις της είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Μια και έχω ελάχιστο χρόνο, θα πω κατευθείαν στα θέματα που με ανησυχούν και με προβληματίζουν. Και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην έκθεση κυρίας Μίλλερ δεν ε, εξηγείται παρκώς ε, το θέμα των φορέων πληρωμής και των αρχών διαχείρισης. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι ο ρόλος των περιφερειών και ο ρόλος ε, στο δεύτερο πυλώνα είναι πολύ σημαντικός να διατηρηθεί. Να κρατήσουμε και τους φόρους ε, πληρωμής και τον εθνικό συντονισμό σίγουρα, αυτά είναι πολύ θετικά, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια το ρόλο που διαδραματίζουν και ανέκαθεν έπαιζαν στο δεύτερο πυλώνα οι περιφέρειες. Και δεν θα πρέπει ε, να συγχαίουμε αυτές τις αρμοδιότητες, γιατί δεν, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια στην πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτι τέτοιο. Κάτι που είπε και η κυρία Εράς. Ε, αυτές οι υπηρεσίες, οι γεωργικές ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ε, νομίζω ότι στην πρόταση της κυρίας Μιλόρ διευρύνεται αυτή η έννοια. Και μάλιστα ε, περιπλέκεται και μια πτυχή αυτής της ε, χρήσιμης ε, συμβουλευτικής υπηρεσίας που θα παίξει κεντρικό ρόλο στο μέλλον. Αλλά καλό θα ήταν να το διευκρινίσουμε. Θα καταθέσω μάλιστα σχετική τροπολογία για να μην καταστήσουμε μη βιώσιμη αυτή την παροχή συμβουλών. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Δεν μπορεί για ένα διοικητικό σφάλμα να περιμένουμε μέχρι και μία τριετία οι γεωργοί για τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Συμφωνώ με τους ελέγχους και συμφωνώ με τα συστήματα, αλλά δεν μπορούμε για ένα μικρό διοικητικό λάθος, που μερικές φορές ε, ε, είναι τελείως άσχετο με τον γεωργό ή δεν φταίει ο ίδιος, να περιμένει δύο και τρία χρόνια για να λάβει τις ενισχύσεις του. Αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε Φυσικά όχι εις βάρος των ελέγχων, ούτε εις βάρος της διαφάνειας. Ευχαριστώ κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο, Άγνιο, ο κύριος Άγνιο πήρε το λόγο. Oh, it's the usual confusion between Agnew and Andrew. Πάλι περτιστήκαμε. Άγνιο και Αντρία δεν ακούγονται καλά τα ονόματα. Αντρία. Πραγματικά Νιώθω απόγνωση αν με μπερδεύετε με τον κύριο Άγνιου. Αντριέ λέγομαι εγώ. Αντριέ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα την κυρία Ούλρη και Μίλλορ ε, για την έκθεσή της αυτή την δύσκολη και κρίσιμη στιγμή και θα είμαι λακωνικός. Εγώ είμαι πραγματικά υπέρ των κοινών κανόνων ε, και για τους ελέγχους και για τις κυρώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να κριτήσουμε και να ενισχύσουμε την κοινή λογική στη νέα μεταρρύθμιση. Και είναι σημαντικό αυτό στην έκθεση. Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό κρίσεων, σίγουρα έχει σχέση με την έκθεση για την κοινή οργάνωση αγοράς. Και συμφωνώ με την έκθεση, με την πρόταση της κυρίας Αράς Καρσία, να είναι σορευτικά τα αποτελέσματα του αποθεματικού των κρίσεων. Και σε ό,τι αφορά την απλούστευση των διαδικασιών, φυσικά θέλουμε απλούστευση και όπως προτείνει και το ελεκτικό συνέδριο, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην απλούστευση και της εφαρμογής. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει να ενισχύσουμε στα σημεία αυτά την έκθεση κυρίας Μίλλερ. Ευχαριστούμε κυρία Αντριέ. Το λόγο κύριος Μπούντα. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιε σύντομε παρατηρήσει για αυτέ τι προτάσει που θεωρούνται είναι πάρα πολύ θετικέ σε σχέση με τον φορέα των αμέσων πληρωμών. Αυτός ο φορέας, αυτός ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί εις των γεωργών, αλλά επίσης θα πρέπει να τους συμβουλεύει όταν έρχεται η ώρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση. Πολλές φορές όμως αυτές οι διαδικασίες είναι γραφειοκρατικές. Είναι δύσκολο να το διεκπαιρεώσουν οι γεωργοί. Χρειάζεται κάποια τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, όσον αφορά την παροχή αυτών των συμβουλών, θα πρέπει αυτή η υπηρεσία να είναι προσβάσιμη εύκολη για τους γεωργούς, ούτως ώστε η διαχείριση της εκμετάλλευσης να γίνεται με τέτοιο τρόπο, που οι Γεωργοί να μην αναγκάζονται να κάνουν λάθη στα διοικητικά και να εφίστανται τις ε, χρηματικές ποινές. Μα είναι και το θέμα της καθυστέρησης το καταβολής των ενισχύσεων στους Γεωργούς. Αν επομένως υπάρχει καθυστέρηση, τι κάνει ο Γεωργός. Οδηγείται στην ε, καταβολή των χρηματικών ποινών. Ναι, αλλά δεν έχει πάρει αυτά που δικαιούται. Δεν θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση ε, να καταλαμβάνει, να καταβάλει τη χρηματική ποινή. Κατάινεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Μίλλερ ε, για την ε, άρτια προετοιμασμένη έκθεσή της. Η έκθεση περιέχει ένα σημαντικό μήνυμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη ακόμη και εν μέσω γεωργική κρίσης και θα πρέπει οι μηχανισμοί διαχείρισης των κρίσεων να μην οδηγήσουν σε ακύρωση των άμεσων ενισχύσεων που είναι απαραίτητε για τους γεωργού. Θα πρέπει ο έλεγχος να ε, βασίζεται στους κινδύνους και οι κυρώσεις ε, να ε, στηρίζονται στην επανάληψη, στην επανειλημμένη διάπραξη λαθών και όχι σε ένα ατύχημα ή σε μια κακοτυχία του Γιώργου. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, είναι σημαντικό να διεκπαιρεώσουμε αυτό το θέμα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία και εύχομαι καλό κουράγιο στην εισηγήτρια για να καταφέρει να διεκπαιρεώσει αυτό το ζήτημα και ελπίζω να συνεργαστούμε με τους και ηγητές για να συμπεριλάβουν αυτά τα τρία σημεία που είναι πολύ σημαντικά και θα επηρεάσουν άμεσα τους γεωργούς. Επαναλαμβάνω, ελπίζω να είμαστε εμπρόθεσμοι ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ, κυρία Μίλλερ. Αυτό που με έπλεξε λίγο στην έκθεσή σα ε, είναι σαν να λέμε ότι το νέο σύστημα το έχουμε ήδη αποδεχτεί. Όμω πρέπει να κάνουμε ε, μια συζήτηση για το κατά πώ θεωρούμε αυτή την με αυτή την ε, τελευταία μεταρρύθμιση. Μην κάνουμε σαν να το δεχτήκαμε ήδη. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Η Κομισιόν κάνει μια πρόταση και ε, προσπαθούμε λιγάκι να τη διορθώσουμε, αλλά γενικώ την δεχόμαστε. Όχι. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ουσιώδη συζήτηση, την οποία ακόμα δεν κάνουμε. Μιλούμε για ελέγχου, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για του ελέγχου. Απ' τη μία ζητούμε λιγότερου αλλά πιο αποτελεσματικού. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε, αν όντω μπορεί να λειτουργήσει. Και επίση πρέπει να προσέξουμε, και αυτό είναι σημαντικό, ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν φτάσει στο ίδιο επίπεδο των ελέγχων. Ε, αυτό είναι το πρώτο βήμα για να μην έχουμε διαφορετικά συστήματα. Και για το παθηματικό για τι κρίσει. Ναι, πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο ταμείο. Πότε θα μπει σε εφαρμογή, πότε θα χρησιμοποιείται. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση που πρέπει επίση να κάνουμε. Θα έχουμε περισσότερε κρίσει, όχι μόνο οικονομικέ. Θα έχουμε και συνεχώ κρίσει, ε, περιβαλλοντικέ και άλλε. Πώ θα τι διαχειριστούμε. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Ερώτημα συγκεκριμένο. Σε ένα σημείο προτείνεται η, τα μέτρα, να υπάρξουν μέτρα ε, ενημερωτικά. Ε, στην Γερμανία αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ. Η CMA καταργήθηκε ε, γιατί είπαμε ότι δεν μπορούμε να ζητούμε τέτοιου είδους πληροφορίες. Εσείς θέλετε να το ξαναεισάγετε στην πρόταση και για, να, για να γίνει τι. Οι καταναλωτές ούτως ή άλλω νιώθουν μια ανασφάλεια. Οπότε εμείς πρέπει ως βουλευτές εδώ να τους ε, διαβεβαιώσουμε. Ε, δεν ξέρω αν ταιριάζει αυτό η υπόλοιπο που κάνετε στον συγκεκριμένο κανονισμό. Ευχαριστώ. Right, Chairman, sorry for, for butting Συγγνώμη για το λάθος προηγουμένως, Πρόεδρε. Πραγματικά πιστεύω ότι ε, σε μένα δώσατε το λόγο. Δεν το έκανα δολίως. Ε, βέβαια. Και κοπίασε για την έκθεση η κυρία Και τελικά ουσιαστικά έχουμε εδώ δύο εκθέσεις. Τα πράγματα είναι απλά στη μία από αυτές. Λέει για το, το ότι μπαίνει σε ένα πρόγραμμα ο, ο Γιωργός και θα πρέπει εκεί να πάρει το χ ποσό. Και θέλουμε να υπάρξει μία αναβολή για δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε είναι δύσκολο αυτό το πρόγραμμα. Τι γίνεται τώρα, υπάρχουν επικονιαστές, υπάρχουν μέλησες τι γίνεται. Κάποιος θα πρέπει να μετρήσει την επίδοση της εκμετάλλευσης. Ακριβώς, όπως θα πρέπει να μετρηθεί το πόσο καθαρό είναι το νερό που χρησιμοποιεί κάποιος γεωργός, κάποιος κτηνοτρόφος, τι γίνεται με την καλομεταχείριση των ζώων, όλα αυτά. Αλλά τι έγινε, μειώθηκαν τα αέρια θερμοκηπίου. Αυτό ποιος θα το μετρήσει. Πώς θα ξέρουμε αυτή την επίδοση. Ναι, κύριε Μιλήρ δεχτήκατε ότι αυτό θα κοστίσει ακόμα και αν γίνεται κάθε δύο χρόνια. Αυτό θα κοστίζει μια περιουσία. Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, κύριε Μαγκίνας, έχω μία ερώτηση, άλλο βέβαια να ευχαριστήσω την Ουλρίκη για τη δουλειά τη. Όσον αφορά αυτή την υπηρεσία παροχή συμβουλών, από τον κανονισμό στρατηγικού σχεδίου να πάει αυτό και να καλυφθεί ε, στον οριζόντιο οικονομισμό. Γιατί γίνεται αυτή η μεταφορά. Καλά τα είπε ο κύριος ε, Άγνιο σε σχέση με το πώς μετράτε η επίδοση σε σχέση με το περιβάλλον. Και να δούμε τι θα μας πει το απόγευμα σχετικά με αυτό το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Μίλλερ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ καλό που έχουμε μια εισηγήτρια που ε, είναι, έχει πραγματικά την οπτική του Γιωργού στο νου τη για την έκθεσή τη Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το κείμενο. Τώρα, το delivery model, ναι, να το συζητήσουμε. Θα το δούμε μάλλον και στα πλαίσια της επόμενης έκθεσης ε, συμφωνούμε κατ' εξαίρεση για το θέμα αυτό, για το τι κάνει η Κομισιόν. Θα πρέπει να δούμε ωστόσο το, ότι αυτή η πολιτική είναι κοινή γεωργική πολιτική. Να μην το ξεχάσουμε αυτό, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αρκετά περήφανοι για την πολιτική αυτή. Υπάρχουν και αντιπροσφορές βεβαίως. Για το σύστημα ελέγχων τώρα, είμαστε σε στενές συζητήσεις, η κυρία Μίλλερ το είπε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με, με την εξίσωση των ε, προτύπων ελέγχων. Αλλά νομίζω ότι στη Γερμανία έχουμε το πρόβλημα ε, με τα τετραγωνικά μέτρα και τις ε, γέες. Ο ο Γιώργο δεν ξέρει. ίσως με το GPS μπορούμε να τα ελέγξουμε, να τα διαχειριστούμε ανά τετραγωνικό μέτρο τι γέε αυτές, Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θέλουμε να ε, μπούμε λίγο στα χωράφια αυτά των γεωργών. Υπάρχουν ε, μέρη όπου δεν ε, υπάρχει χορτάρι πια, δεν φυτρώνει πια χορτάρι. Θα πρέπει ίσως να μην καταργήσουμε τελείως τα πρότυπα ελέγχων και επίση ε, στα σημεία που είπε η, ε, η ότι θέλει να κάνει τροποποίηση για να βελτιωθεί, θα πρέπει όντω να έχουμε υπόψη μα πάντα τη βελτίωση υπέρ του γεωργού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια για την εξαιρετική της έκθεση. Το βασικό δίλημα είναι αυτό αυτή, αυτό το σκεπτικό, αν θα το ακολουθήσουμε ή αν θα ακολουθήσουμε κάτι άλλο. Ε, πολλοί έχουν ε, ξανασυζητήσει για το θέμα αυτό, για την ε, σύσταση του κυρίου Ντόρφμαν και συζητήσαμε και συμμετείχαμε ενεργά στην αντιπαράθεση για την έκθεση αυτή και τις προτάσεις της Κομισιόν όντως θα πρέπει να τις βελτιώσουμε γιατί αλλιώς ο γεωργικός τομέας πραγματικά θα πληγεί. Την έκθεση λοιπόν της συναδέλφου την υποστηρίζω, ας πούμε την διετή υποβολή εκθέσεων. Κατά την απόψή μου θα μπορούσαμε να την κάνουμε και τρία χρόνια. Νομίζω ότι η Κομισιόν στα κείμενα θα πρέπει ξεκάθαρα να προτείνει αυτό που θέλει να προτείνει και εμείς να αποφασίσουμε αν μας ικανοποιεί ή όχι. Τα, ε, τα δύο χρόνια τουλάχιστον για μεταβατική περίοδο πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και στο, το 2023 θα μπορεί αυτή η πολιτική να εφαρμοστεί. Τώρα, σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα πρέπει ε, να έχουμε υπόψη και τις ε, καταστροφές που μπορεί να συμβούν ή τις κρίσεις. Ε, ας πούμε, αν κάποιος χάσει ένα μέλος της οικογένειάς του που δουλεύει στην οικογενειακή φάρμα, εκεί θα πρέπει να έχουμε προβλέψει. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδου στήριξη. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης ανταλλαγή ε, τεχνογνωσίας και ψηφιοποίηση για να μην είναι δύσκολο όλα αυτά για τον Γιώργο. Κυρία Ντελέ, ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν ευχαριστήσω την κυρία Μίλλερ για το έργο της και να επανέλθω στο ζήτημα του αποθεματικού κρίσεων. Να έχουμε ένα αποθεματικό κρίσεων με προπολογισμό 400 εκατομμύρια ενώ έχουμε πρόσφατες αναμνήσεις από το πόσο κόστησε η γαλακτοκομική κρίση, τι να πω, είναι πενιχρός ο προπολογισμό καθόλου φιλόδοξη αυτή η πρόταση των 300 εκατομμύριων για το αποθεματικό κρίσεων. Επίσης, ε, συμφωνώ να αντικαταστήσουμε τις εφαρμοστικές πράξεις από τις κατεξιοδότηση πράξεις. Θα πρέπει να κρατήσουμε κάποιο κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εφαρμογή της κοινή γεωρικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Δεκάστρο. Η έκθεση της συναδελφού Μιλέρ πάει στη σωστή κατεύθυνση για αυτές τις κοινέ ε, αρχές και για τις ε, κυρώσεις όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με την αιρεσιμότητα. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι κοινοί κανόνες για έλεγχο, διοικητικές κυρώσεις και ανάκτηση των αχρεωστήτων. Επομένω θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδου κοινή διαχείριση, διακυβέρνηση, ασφάλεια δικαίου, περισσότερη για τους γεωργού μας. Όσον αφορά τώρα το αποθεματικό, θα συνεργαστούμε με τον κύριο Σάντος, ώστε αυτό το, αυτά τα 400 ε, εκατομμύρια ω πρικοδότηση να αυξηθούν. Γιατί χρειάζεται ε, στην περίπτωση κρίσης διαφορετικά κριτήρια μέτρησης των επιδόσεων και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον οριζόντιο κανονισμό. Κλονέκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπράβο στην Ουλρίγε για τις ε, προτάσεις της που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Συμφωνώ με πολλά που έχει το κείμενό της, κυρίως για απλούστευση, μείωση της γραφειοκρατίας, γιατί η Κομισιόν δεν μας καλύπτει αρκετά με τις προτάσεις. Τώρα, όσον αφορά το αποθεματικό κρίση. θα πρέπει να αφορά τη γεωργία. Θα πρέπει να προοικοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό, όπως είπε και η Αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε θα πρέπει να τροφοδοτείται με φρέσκα κεφάλαια τα χρήματα του πρώτου πυλώνα. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τις κρίσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε το κατάλογο των αγοριτών για το θέμα αυτό. Δεν βλέπω να ζητά άλλος κανείς το λόγο. Οπότε θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον κύριο Μέγκελε, να σχολιάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μίλλερ για το σχέδιο έκθεσης που υπέβαλε και ε, να την επενέσω για το διαλεκτικό της πνεύμα και την προθυμία της για συζήτηση. Είχαμε ήδη πολλές συναντήσεις ε, με την εισηγήτρια, όπου παρουσιάσαμε πολύ πιο διεξοδικά τον κανονισμό. Είναι πολύ καλή βάση και για την περαιτέρω διαδικασία και συνεργασία. Ε, αυτό το, αυτός ο κανονισμός αφορά τη διαχείριση της ΚΑΠ. Ε, διαχείριση από διοικητικούς φορείς, από τα κράτη-μέλη, ε, με ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή. Οπότε ο κανονισμός αυτός είναι απαραίτητο, παρόλο που είναι αρκετά τεχνικός και περίπλοκος. Μιλούμε για, τη, για δημοσιονομικές διαδικασίες και για αποφάσεις ε, σε αυτό το πλαίσιο. Εξού και η αλλαγή που προτείναμε, οι ελάχιστε αλλαγές που προτείναμε στον κανονισμό, γιατί ο κανονισμό αυτό μέχρι στιγμή εφαρμόζεται και ήδη λειτουργεί. Επισημάναμε το χαμηλό ποσοστό σφάλματο, που είναι συναφές με την καλή λειτουργία του κανονισμού. Και γι' αυτό περιορίσαμε το έργο μα σε κάποιε προσαρμογέ του κειμένου στη νέα πολιτική που έχει προταθεί και που περιχαρακώνεται στον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάτε. Η πρόταση αυτή ουσιαστικά αξιοποιεί τα ήδη υπάρχοντα. Για τα μέτρα πληροφόρηση, για παράδειγμα, δεν αλλάζουμε τίποτα. Απλώς αλλάζουμε το, το σημείο που αναφέρεται η διάταξη. Παλιά ήταν στο 40 και, τώρα είναι στα πρώτα 10 άρθρα. Ένα άρθρο που ήδη υπήρχε, που δεν έχει καμία θέση με το CMR και καμία αλλαγή στα μέχρι τώρα ισχύοντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους παρατηρήσεις, θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις. Καταρχήν, αναφέρονται κάποιοι ορισμοί που αναφέρονται και στο κανονισμό περί κοινών διατάξεων, το CPR. Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων εξακολουθεί να εδράζεται στην παλιά προσέγγιση περί συμμόρφωσης. Οπότε δεν νομίζω ότι ευσταθούν αυτές οι μνήες ούτε συνάδουν με τον οριζόντιο κανονισμό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φορείς διαχείρισης, οι αρχές διαχείρισης, άλλαξε η σειρά των άρθρων. Και αυτό είναι συζητήσιμο. Και το κατά πόσο είναι λογικό. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε στη συνέχεια ίσως. Μία αλλαγή όμως μας ανησυχεί και μας προβληματίζει, γιατί δίνεται στους συντονιστικούς φορείς σημαντικό διαχειριστικό ρόλο. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, οι συντονιστικοί φορείς στα κράτη-μέλη υπάρχουν μόνο σε χώρες που υπάρχουν περισσότεροι φορεί πληρωμής και ουσιαστικά έχουν συντονιστικό ρόλο. Δεν έχουν ξεχωριστό ρόλο, ένα ιδιαίτερο ρόλο πολιτικής. Και αυτό φαίνεται ότι θέλετε, γιατί αυτό κατάλαβα από τη συζήτηση, ότι θέλετε να προσδιορίσετε με σαφήνεια τις περιφερειακές αρμοδιότητες στην πολιτική. Και αυτό που κάνετε εδώ είναι να μεταφέρετε αρμοδιότητες και ευθύνε σε κεντρικό επίπεδο. Σε ένα φορέα που ουδέποτε δεν είχε εκτελεστική αρμοδιότητα ή ουδέποτε δεν είχε τόσο ουσιαστικό ρόλο. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Επίσης, οι ε, αρχές διαχείρισης ε, και τα, οι γεωργικές ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες πέρασαν από τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια στον οριζόντιο κανονισμό. Αυτό δεν είναι τραγικό, αλλά είναι κάπως προβληματικό, γιατί αυτές οι διατάξεις ε, είναι τμήμα του πολιτικού πλαισίου και έχουν σωστή θέση στον κανονισμό περί στρατηγικών σχεδίων και όχι στον οριζόντιο κανονισμό. Κάτι που αναφέρθηκε από πολλούς ε, ε, ομιλητές, ό,τι αφορά την ετήσια ε, καθάριση, ό,τι αφορά τις επιδόσεις. Αυτό μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο. Αυτή η καθάριση των επιδόσεων είναι μια διαδικασία που σχετίζεται με τη, τις δηλώσεις που έχουν ετήσιο χαρακτήρα. Αν κάνετε διαιτή το χαρακτήρα, θα δημιουργήσει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ε, δήλωση αξιοπιστίας και δεν συνάδει ούτε με τον δημοσιονομικό κανονισμό που μιλάει για το πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η δήλωση αξιοπιστίας. Η υποβολή δηλώσεων. Γι' αυτό ξανασκεφτείτε παρακαλώ τις αλλαγές που προτείνετε. Επίσης, ε, μερικές φορές αναφέρθηκαν, ε, αναφέρθηκε το θέμα του αποθεματικού, του γεωργικού αποθεματικού. Και προτάθηκαν κάποιες μη ρεαλιστικέ ιδέε. Γιατί είπατε να καταργηθεί το τρέχον αποθεματικό κρίσεων που κρίθηκε αναποτελεσματικό. Δεν λειτουργήσε γιατί δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί. Οπότε αυτό που προτείνουμε είναι ένα γεωργικό αποθεματικό που είναι απλώς μία δημοσιονομική γραμμή. Ένα άρθρο στον προϋπολογισμό που συνδυάζει όλα τα σημεία που, όλα τα, τα συγγνώμη, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν κρίσει ή να διαχειριστούν την αγορά. Τώρα, ποιο θα είναι το ποσό προπολογισμό αυτού του γεωργικού αποθεματικού είναι ζήτημα πολιτική λύση. Εμεί προτείναμε τουλάχιστον 400 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι η αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή μπορεί να αυξήσει τον προπολογισμό. Οπότε, όποιο και είναι ο προπολογισμό του γεωργικού ταμείου, αν κρυθεί ε, έλλειπης ή αναποτελεσματικός, δεν αποκλείεται να ε, αυξηθεί ο προπολογισμό του γεωργικού αποθεματικού. Αλλά δεν υπάρχει λόγο να περάσουμε από το γεωργικό αποθεματικό σε ένα αποθεματικό μέτρα αγοράς κάποια θέσεις γιατί ούτω ή άλλω τα μέτρα αγορά κάποια θέση στον προπολογισμό θα πρέπει να έχουν. Οπότε προ τι η πρότασή σα για το αποθεματικό κρίσιο, που ήταν αναποτελεσματικό. Σε τελική ανάλυση το ζήτημα είναι οικονομικό. Πόσα κονδύλια θα πρέπει να αφιερωθούν ή να περιλουθούν στον προπολογισμό για μέτρα αγοράς. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι γεωργικό, αποθεματικό, αποθεματικό κρίσεων ή σε ποιε δημοσιονομικέ γραμμέ θα συμπεριληφθούν. Αυτή η συζήτηση μα αποσπά την προσοχή μα από το ουσιώδη. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ανώτατων ορίων, ίσω και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί, γιατί τα οικονομικά αυτά ανώτατα όρια είναι απαραίτητα για τη δημοσιονομική διαχείριση. Γιατί θέλετε να καταργηθούν. Και στο άρθρο 45 του κανονισμού, ε, το όρ το αντικαταστήσει από το end. Αυτή η αλλαγή μπορεί να είναι σοβαρή, είναι δυνητικά σοβαρή, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να τη δούμε στα πλαίσια μιας γενικής βελτίωσης του άρθρου 35 και μιας διευκρίνησης των διατάξεων που για μερικούς φαίνονται ασαφείς, γιατί ήδη έχουμε συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό και ίσως βρούμε κάποια λύση για το άρθρο 35. Επίσης, είπατε, θέλετε να αποκλείσετε περισσότερους γεωργούς από τα πρόστιμα και τις κυρώσεις. Αυτό είναι νέο θέμα αιρεσιμότητας, αλλά ίσως έτσι οδηγηθούμε σε ευρύτερες εξαιρέσεις από τις ισχύουσε. γιατί οι παρούσες εξαιρέσεις αφορούν μόνο την οικολογικοποίηση. Αλλά τώρα θέλετε να εξαιρέσετε κάποιους γεωργούς και από την πολλαπλή συμμόρφωση αμέσως, κάτι που δεν συνάδει με την αύξηση των περιβαλλοντικών μας φιλοδοξιών δεν θα πω τίποτα για τις εφαρμοστικές ή καταξιοδότηση πράξεις, γιατί αυτό είναι ένα από τα δύσκολα θεσμικά ζητήματα που ίσως συζητηθούν στον τελευταίο τριμερή διάλογο, που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Γιατί αυτό είναι θέμα Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Είναι θεσμικό περισσότερο ζήτημα. Και ένα λεπτό ακόμη επιτρέψτε μου να μιλήσω για κάποια άλλα ζητήματα. Ανωτέρα βία διαγράψαμε αυτή τη διαδικασία γιατί σε ένα σύστημα που έχει μεγαλύτερη επικορικότητα για τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει ε, να νομοθετούμε εμείς με μεγάλες λεπτομέρειες. Και αν θέλετε να ε, επαναφέρουμε την κατάσταση ε, θανάτου του Γεωργού ή σοβαρού τυχήματο που είναι λόγια νοτέρας βίας, αν θέλετε να το επαναφέρουμε δεν είναι πρόβλημα. κυρία Χόιμπουχ αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή πολιτική. Εγώ θα ήμουν υπέρ της σχετικής συζήτησης στα πλαίσια του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια, γιατί εκεί είναι που μιλούμε για τις πολιτικές. Ο οριζόντιος κανονισμός, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένας κανονισμός διαχειριστικός, είναι τεχνικός, αφορά τους θεσμούς, τους φορείς, τις διαδικασίες και όχι την ουσία της πολιτικής και κυρίως όχι την εξωτερική πολιτική. Και θα ήταν λάθος να φέρουμε ένα τέτοιο θέμα στον οριζόντιο κανονισμό. Να το συζητήσουμε μεν, αλλά στα πλαίσια του κανονισμού για στρατηγικά σχέδια. Τώρα, νησιν 2 ή νησιν 3. Στο παρελθόν είχαμε νησιν 2, που σημαίνει ότι η αγροτική ανάπτυξη... Ε, για την αγροτική ανάπτυξη τα κράτη-μέλη έχουν δύο χρόνια για να δαπανίσουν τα κονδύλια. Δύο χρόνια μετά την δέσμευση που αναλύθηκε. Και το 2013 το νησιν 2 έγινε νησιν 3 γιατί σκεφτήκαμε ότι δίνοντας τα κράτη-μέλη περισσότερο χρόνο, ίσως μειώνουν το σφάλ, τα, τα ραλ, τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, τα, ανα, ε, τα χρησιμοποιητά κονδύλια δηλαδή. Γιατί μερικές φορές ε, οι καθυστερημένοι λογαριασμοί και απλήρωτοι λογαριασμοί μαζεύονται σε χιονοστιβάδα. Και είδαμε ότι το νησιν 3 δεν λειτουργήσε. Όσο περισσότερο χρόνο δίνουμε στις αρμόδιες αρχές, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζονται και τον διεκδικούν. Οπότε σκεφτήκαμε ότι έχει νόημα να επιστρέψουμε, να επανέλθουμε στον ΙΣΙΝ γιατί ίσω μία μικρή πίεση χρόνου αναγκάζει τα κράτη-μέλη να εντείνουν τι προσπάθειέ του και να επιταχύνουν την απορρόφηση, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο τη δημοσιονομική διαχείριση. Κύριε Αγγιλέρα, αναφερθήκατε στου φορεί πληρωμή και τη διευκρίνηση του ρόλου του, όπω είπα και στην αρχή. Εμεί δεν αλλάξαμε και πολλά στο σημείο αυτό. Ο ρόλος των φορέων πληρωμής είναι καθαρός και εξάστερος και ανέκαθεν ε, είχε γίνει αντιληπτό σωστά. Μικρές προσαρμογές κάναμε στη νέα πολιτική και μάλιστα το συζητήσαμε και στο δίκτυο φορέων πληρωμής. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε περαιτέρω για να μου επισημάνετε κάποια τεχνικά σημεία που κατά τη γνώμη σας είναι ασαφή και χρήζουν διευκρίνησης. Και αναφέρθηκα και στα μέτρα πληροφόρησης. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σχέση με την παρούσα κατάσταση και προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτού του εντατικού διαλόγου για να φέρουμε αυτή τη διαδικασία σε αίσιο πέρα, σε συνεργασία με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μέγκελε. Ο κύριος Άγνιος ζήτησε το λόγο για συμπληρωματικές ερωτήσεις. This is a order. Για διαδικαστικό θέλω πρόεδρε. Για να θέσω το εξής. Άκουσα δύο αγγλικές, δύο αγγλικές λέξεις διαιτές και διαιτές. Ναι, αλλά τι είναι αυτό, κάθε έξι μήνες ή κάθε δύο χρόνια. Biannual και biennial. Μην τα μπερδεύετε, δεν ξέρω, δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί αν δεν γίνει σωστά η διάκριση, βλέπω να έχουμε πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, οπότε ξαναδίνουμε το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρεμβάσεις. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι όντως χρειαζόμαστε μια καλή βάση για να παραμείνουμε σε συζήτηση και να εξαντλήσουμε τα θέματα που παραμένουν εκκρεμή. Φυσικά εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, αλλά προσπαθούμε όλες αυτές να τις συγκεράσουμε στην έκθεση. Ε, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, βεβαίω δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα επιμέρου ερωτήματα και να σχολιάσω τι ε, παρεμβάσει. Απλώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, να συνεργαστώ με του ε, σκιώδε ηγητέ, γιατί όντω επί τη ουσία πρέπει να επιφέρουμε απλουστεύσει στη διοικητική διαχείριση για τους γεωργούς και χαίρομαι βεβαίως που θα λάβω τις τροπολογίες των συναδέλφων σίγουρα και με τους εισηγητές των άλλων δύο κανονισμών θα είμαστε σε στενή συνεργασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τους, ε, τον οριζόντιο ε, κανονισμό ο οποίος ασχολείται και με, την, ε, και με τη ΣΚΟΑ και με τα στρατηγικά σχέδια. Ευχαριστώ λοιπόν και χαίρομαι για την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Μέχρι 3 Δεκεμβρίου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας στις 3 το μεσημέρι. 3 Δεκεμβρίου 3 το μεσημέρι λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες και να περάσουμε ευχαριστώντας την κυρία Μίλλερ και του συναδέλφου που έλαβαν μέρο στη συζήτηση στο επόμενο θέμα. Και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι σας έχουμε διαβιβάσει μία επιστολή που μου έστειλε ο πρόεδρος Ταγιάννη. Στην επιστολή του κυρίου Ταγιάννη, του πρόεδρου, αναφέρεται ένα ζήτημα για τα τομεακά προγράμματα και μιλά για το άρθρο 59α και την παραπομπή στην Ολομέλεια και το άρθρο 69 για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα γιατί θα μας αναγκάσει να επιταχύνουμε αισθητά τις εργασίες μας. Θα το πούμε και στους συντονιστές, αλλά θα ήθελα να σας επισημάνω την αποστολή αυτής της επιστολής από τον Πρόεδρο Ταγιάννη. Και να περάσουμε στο επόμενο τώρα σημείο τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη στήριξη στρατηγικών σχεδίων που θα καταρτιστούν από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτά τα περιβόητα στρατηγικά σχέδια κοινή γεωργικής πολιτικής που θα χρηματοδοτηθούν, που θα εμπίπτουν στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα και εμείς είμαστε αρμόδιοι επί τη ουσία, αλλά γνωμοδότηση έχουν δώσει διάφορε επιτροπέ μεταξύ άλλων και Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μάλιστα, μερικοί από τους συντάκτες γνωμοδότης είναι και μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Και ως μέλη και άλλων επιτροπών κατέρθησαν τις γνωμοδοτήσεις για τις άλλες επιτροπές. Θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ρανς Γκαρσία, και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Κυρία Γκαρσία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βέβαια γιατί είχαμε πολύ στενή συνεργασία από την αρχή και είχαμε επαφή αμέσως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις εργασίες, γιατί το πρόβλημά μας ήταν ο ελάχιστος χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Πάντως ήταν πολύ πρόθυμη για συζήτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέσω, αλλά και το Συμβούλιο, γιατί και τα μέλη του Συμβουλίου προσπάθησαν και εξέφρασαν αμέσω τις απόψεις τους για το έγγραφο. Και τα μέλη των ομάδων πίεση ε, ε, με συνάντησαν πολλές φορές. Έχουν έρθει από συνδικάτα, από συνεταιρισμούς, από τον κλάδο. Γενικώ όλοι έσπευσαν να ασχοληθούν με τις συζητήσεις. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες του εγγράφου. Καταρχήν, έτοιμα ενός επαρκούς προϋπολογισμού για την κοινή πολιτική. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα Συνεχίζονται οι συζητήσει Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που έχει μεταρρύθμιση της κοινή γεωρική πολιτικής. Το δεύτερο σημείο είναι οι προθεσμίε. Θέλουμε αναβολή της εφαρμογή των ε, στρατηγικών σχεδίων μέχρι την έγκρισή τους και την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εγκρίνουν ε, τα σχέδια αυτά. Και βάζω το 2023 σήμερα ημερομηνία, γιατί είναι αρκετά περίπλοκα αυτά τα στρατηγικά σχέδια. Θέλω να δώσουμε χρόνο στα κράτη-μέλη, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνο να καθυστερήσουν οι ενισχύσει προς τους γεωργούς. Και τρίτο στοιχείο που ζητούμε είναι η ενίσχυση των κοινών στοιχείων της κοινή γεωργική πολιτικής. Όπω είπαμε στη συζήτηση που είχαμε πριν συντάξω το σχέδιο Έκθεση, ένα από τα βασικά μελήματά μα ήταν να έχουμε πολλά κοινά στοιχεία στα στρατηγικά σχέδια. Και ακριβώ λόγω αυτών των κοινών στοιχείων από την αρχή να εξακολουθήσουμε και στο μέρο να διαφυλάσσουμε τον κοινό χαρακτήρα της αγροτικής μας πολιτικής. Χρειάστηκε να καταλήξουμε σε μια σειρά στόχων, γενικών στόχων και ειδικών στόχων, καθώς και στη θέσπιση διαφόρων δικτών. Σε ό,τι αφορά τους στόχους, με την ε, εισαγωγή των γενικών στόχων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξασφάλιση κατάλληλου ε, γεωρικού εισοδήματος και αξιοπρεπής ε, και αξιοπρεπών τιμών για τους καταναλωτές είναι το βασικό σύνθημα, η βασική αποδός και εξασφάλιση του γεωρικού εισοδήματος και προσιτές τιμές για τους καταναλωτές. Βλέποντας τις διεθνείς ε, συνθήκες και τις δικές μας επιλογές, βλέπουμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα κατάλληλο γεωρικό εισόδημα. Και επίσης για, τα καταναλωτό, για τους καταναλωτές θα πρέπει να μειώνεται το τμήμα του προϋπολογισμού του νοικοκυριού που αφιερώνεται στη διατροφή. Και πραγματικά έχει μειωθεί ε, το κονδύλι που αφιερώνει οι καταναλωτές στη διατροφή. Και αυτό είναι σημαντικό στόχος και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί στόχο και στο μέλλον. Επίσης, ε, να περιοριστεί η σπατάλη τροφίμων. Αλλά δεν έχει μεγάλη συνέπεια για τη γεωργία. Συμφωνώ να περιοριστεί η σπατάλη τροφίμων, αλλά δεν αφορά αυτό τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Επίσης, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της γυναίκας στη γεωργική οικονομία. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγροτική οικονομία είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο λόγω δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να συμβάλλουν και οι γυναίκες για να καταπολεμηθεί η απερίμωση της υπαίθρου και να αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές απειλές. Γιατί ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γυράσκει και οι νέες γυναίκες δεν έχουν ε, παιδιά για να εξασφαλιστεί η ηλικιακή ανανέωση του πληθυσμού. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες, περιλαμβάνω και νέους δείκτες για τις γυναίκες, ε, συμβάλλουν ε, τα δάση στην εξυγίαση του αέρα και την ε, επίτευξη νέων αγορών. Και επίσης ε, δεν θέλουμε εξοδότηση πράξης να περιλαμβάνει νέους δείκτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση. Η σημαντικότερη συζήτηση θα είναι για τους ορισμούς. Μόνιμα βοσκοτόπια, νέοι, νεαροί γεωργοί. Ε, η έννοια του γνήσιου γεωργού ή του ενεργού γεωργού. Για το γνήσιο Γεωργό, τον ενεργό Γεωργό, άκουσα τις απόψεις σας, άκουσα τις θέσεις των κρατών μελών, άκουσα τα λόμπι και ε, θα είναι σφοδρή η συζήτηση που θα έχουμε για την έννοια του γνήσιου Γεωργού. Εγώ τροποποιώ την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνδέω τον ορισμό του γνήσιου Γεωργού με την γεωργική δραστηριότητα και την προστασία του οικογενειακού γεωργικού μοντέλου και του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί ώστε ο ορισμός του γνήσιου γεωργού να είναι όσο πιο ευρύς γίνεται για να τύχει τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη στην Επιτροπή μας. Ό,τι αφορά τα μόνιμα βοσκοτόπια. Συμπεριλαμβάνω εδώ τον ορισμό που υπάρχει ήδη στον κανονισμό Omnibus για να συμπεριληφθούν και τα ειδικά ε, ισπανικά βοσκοτόπια, τα DESAS, που περιλαμβάνουν και χαμηλή δασική βλάστηση. Σε ό,τι αφορά τους νέους αγρότες, υπάρχει δυνατότητα κάποια χώρα μετά από μελέτη να κρίνει ότι χρειάζεται διεύρυνση του ηλικιακού φάσματος, να φτάσουμε στα 40-45 χρόνια. Γιατί όχι. Γιατί πραγματικά ο μέσος, η μέση ηλικία του, του Γεωργού σε πολλά κράτη-μέλη είναι αρκετά υψηλή. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ηλικία για τον ορισμό του νέου Γεωργού. Γιατί ίσως κάποιες χώρες το κρίνουν απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά τους νέους Γεωργούς, τους νέους ερχόμενους, ε, αλλά περιλαμβάνω έναν ορισμό σε σχέση με τις, βοηθήσεις, με τις, βοή, ενισχύσεις και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ηλικιακή ανανέωση και στην καταπολέμηση της απερίμωσης της υπαίθρου. Επίσης προτείνω ε, κάποιες ε, παρεμβάσεις για τις άμεσες ενισχύσεις. Προτείνω ε, βασική ενίσχυση για τη βιωσιμότητα και επίσης τουλάχιστον 70% των άμεσων ενισχύσεων να συμβάλλουν στη σταθερότητα των γεωργικών εισοδημάτων και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά μέτρα της έκθεσής μου σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια, το κάπινγκ που λέμε. Και αυτό προβληματίζει πολλούς συναδέλφους. Κατά τη γνώμη μου, να είναι υποχρεωτικό το κάπινγκ για τα κράτη-μέλη και να υπάρχει δυνατότητα ε, θέσπισης ενός νέου κατοφλίου που δεν θα είναι ποτέ κατώτερο από 1.000 ευρώ μετά την έκπτωση των μισθών, ε, τις ενισχύσεις για, το, για την οικολογικοποίηση και τις ενισχύσεις για τους νέους γεωργούς. Πολλές διοικήσεις μου έκαναν παράπονα και πολλοί γεωργικοί συνεταιρισμοί γιατί κρίνουν ότι η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διαφορετικές παραγωγικές δομές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές των κρατών μελών κατά τη θέσπιση του κάπινγκ. Και γι' αυτό εγώ αφήνω κάποιο περιθώριο επικουρικότητα στα κράτη-μέλη. Πάντως, ε, περιμένω τις απόψεις και με διαλλακτική. ό,τι αφορά την α, αναδιανεμητική εισφορά, 25% τη βασική ενίσχυση στο εισόδημα τη βιωσιμότητας και τουλάχιστον ένα ανώτατο όριο 30 εκτάρια ή αντίστοιχο με το μέσο όρο των γεωρικών εκμεταλλεύσεων των κρατών μελών. Επίσης με κάποια άλλα κριτήρια για να εξασφαλίσω μια δίκαιη κατανομή, ακριβώς δίκαιη κατανομή αυτής της πληρωμής. Ό,τι αφορά το οικολογικό σύστημα, προτείνω οι, οι αυτού του νέου μηχανισμού να είναι διαφορετικές ή συμπληρωματικές σε αυτές που αφορούν τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και τα κλιματικά μέτρα. Το οικολογικό σύστημα είναι ετήσιο, ενώ τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα είναι πολυετή. Θα μπορούσαν λοιπόν τα δύο συστήματα να είναι συμπληρωματικά. Θα μου πείτε και εσείς τι γνώμη έχετε. Πάντως πιστεύω ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Επίση, τη δυνατότητα στα πλαίσια των οικολογικών συστημάτων, των οικολογικών συνιστοσών, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάποια ευνοϊκά αγιορικά συστήματα που ήδη πληρούν υψηλέ περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ. Για παράδειγμα, εκτατική κτηνοτροφία. Η εκτατική κτηνοτροφία έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην Ήπεθρο, ιδιαίτερα στι ορεινέ περιοχές. Και δεν είχε αναγνωριστεί ποτέ αυτό. Θα θυμάστε ε, την έκθεση για τα εγωπρόβατα. Εκεί θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε το έργο των εγωπροβατοτρόφων. Σε ό,τι αφορά την αρεσιμότητα. Είναι πολύ ενισχυμένη. Καταργείται το θέμα της βιωσιμότητας των θρεπτικών ουσιών στα πλαίσια των βέλτιστων γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών. Γιατί έλαβα υπόψη τις δυσκολίες που ίσως δημιουργήσει η εφαρμογή του μέτρου για ζώνες που δεν έχουν καν ευρυζωνικό διαδίκτυο. Γι' αυτό προτείνω η βιωσιμότητα των ε, θρεπτικών ουσιών να συμπεριληφθεί στα συστήματα αξιολόγησης. Επίσης, διατηρώ τους ισχύοντες κανόνες για τις ισοδυναμίες ε, σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα. Σε ό,τι αφορά τη βιολογική γεωργία και τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ, θα πρέπει να εξαιρούνται από τι βέλτιστες γεωργικέ και περιβαλλοντικέ πρακτικέ που συνδέονται με την ε, οικολογικοποίηση, ε, γιατί έχουν ιδιαίτερότητε Και η βιολογική γεωργία ήδη εκφίσωση είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά και οι εξόχω απόκεντρε περιοχέ έχουν διαφορετικέ πολύ διαφορετικές περιστάσεις και συνθήκες από τις υπόλοιπες περιοχές. Σε ό,τι αφορά τις γεωργικές πρακτικές, επαναφέρω κάποια κεντρικά σημεία, ε, επίκαιρε ε, περιβαλλοντικές πρακτικές και επίσης ε, το κατόφλι διαφοροποίησης 5% για μόνιμους βοσκοτόπους, δυνατότητα πρωτεϊνούχων καλλιεργιών σε, σε περιοχές αγρανάπαυσης και επίσης ε, η εξαίρεση των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων κάτω των 10 εκταρίων. Σε ό,τι αφορά τους νέους γεωργούς, ε, δεν θέλουμε παλιδρόμηση για να μην περιοριστούν τα κονδύλια για τους νέους γεωργούς. Γιατί σήμερα, αν έχουμε υπερβολικές δαπάνες για τους νέους γεωργούς, χάνει το κράτος μέλος. Οπότε περιλαμβάνω αυτή την ρήτρα της μη υπαναχώρησης. Επίσης, ε, περνάμε από 5 σε 7 χρόνια για τη διάρκεια αυτής της ενίσχυσης. Ό,τι αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, τις κρατώ στο επίπεδο που ε, ισχύει τώρα και 2% επιπλέον προτείνω για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Σε ό,τι αφορά το εθνικό αποθεματικό, βάζω ένα ανώτατο όριο, 3% για, τις, για τα δικαιώματα πληρωμής, όπως ισχύει και τώρα. Και σε ό,τι αφορά τις ε, τομεακές παρεμβάσεις, περιλαμβάνω τη ρήτρα που εξασφαλίζει την απαραίτητη μετάβαση στο νέο στα νέα προγράμματα, από τα παρόντα στα νέα. Σε ό,τι αφορά τους άλλους τομείς, το, το επεκτείνω και σε άλλα προϊόντα, όπως πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Και επίσης ε, τη δυνατότητα εκπόνηση όχι μόνο λειτουργικών προγραμμάτων, αλλά και εθνικών προγραμμάτων στήριξης, όπως υπάρχουν για το κρασί ή για τη μελισσοκομεία. Σε ό,τι αφορά τη μελισσοκομεία, από 50% περνάμε στο 75% ποσοστό συγχρηματοδότησης. Είχαμε πει στην προηγούμενη συζήτηση ότι με την αύξηση του προπολογισμού για τη μελισσοκομεία είναι λογικό να αυξήσουμε και το ποσοστό συγχρηματοδότηση. Για τα οποροκυπευτικά προτείνω πιο ρεαλιστική περιβαλλοντική φιλοδοξία και μιλώ για 10% των λειτουργικών κονδύλιων που θα πρέπει υποχρεωτικά να αφιερώνονται σε περιβαλλοντικά μέτρα λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι διαγράφεται η επιλογή δύο μέτρων ως εναλλακτική για το 100%. Οπότε δεν δικαιώνομαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ούτε δικαιώνω τον κλάδο. Υιοθετώ μια χρυσή τομή, μια μέση λύση. Και προτείνω και νέα κίνητρα για να ενισχύσουμε την οργάνωση σε οργανώσεις παραγωγών και σε ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Θέλουμε να υπάρχει μια συγκέντρωση της προσφοράς και παροτρύνουμε τους οργανισμούς, τους ε, γεωργούς να οργανωθούν. Σε ό,τι αφορά για το κρασί, ε, υπέρ των επενδύσεων στην καινοτομία ευνοώντας όχι μόνο τις μεγάλες αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί και οι, μεγάλε, οι μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως κάνουν επενδύσεις σε καινοτομίες που στη συνέχεια ωφελούν το σύνολο του κλάδου. ό,τι αφορά τη γεωργική ανάπτυξη, την ε, αγροτική ανάπτυξη, εκεί τα φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα προτείνω να είναι υποχρεωτικά σε όλη την επικράτεια των κρατών μελών. Και πιστεύω ότι αυτές οι ενισχύσεις θα πρέπει να δίνονται όχι μόνο σαν αντιστάθμιση του διαφυγόντος κέρδους, αλλά και ως κίνητρο προτείνω διαγραφή στην πρόσβαση στις ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία και τους γνήσιους γεωργούς ως τους μοναδικούς δικαιούχους. Επίσης, προτιμώ να δώσουμε έφεση στους ενεργούς γεωργούς. Σε ό,τι αφορά τις ζώνες με φυσικές μειονεξίες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό για το 30% των ενισχύσεων. Οπότε, αν οι ενισχύσεις αυτές, αν για την επικράτεια ε, θα πρέπει το 30% ε, να δοθεί σε περιβαλλοντικές και κλιματικές αλλαγές, να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα αυτών των περιοχών με ιδιαίτερες μειονεξίες. Και να ληφθεί υπόψη ο ο ρόλος των ε, περιοχών αυτών στην ε, διαφύλαξη της βιοπικιλότητας. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, τις μεγάλες επενδύσεις της Γεωργία, σε ό,τι αφορά τους νέους γεωργούς, το συνδέω με τους νέους ερχόμενους και εκεί περιλαμβάνω και τη βοήθεια στην εγκατάσταση των νέων γεωργών. Διαφυλάσσω την βοήθεια στους στους γεωργούς που μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους σε νέους γεωργούς και επίσης ο γεωργός που φτάνει στην συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχει κάποια κίνητρα για να μεταβιβάζει την εκμετάλλευσή του σε κάποιον άλλο γεωργό εκτινοτρόφο που θα κρατήσει την γεωργία στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για τα ημείωση του κινδύνου, ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συστημάτων που να καλύπτουν πολλούς κινδύνους ή ταμεία συνεταιρισμών ή οργανώσεων παραγωγών. Σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή ε, γνώσεων, Αυξάνεται η συγχρηματοδότηση από το 75% στο 100% για μέτρα που στόχο έχουν την ανταλλαγή γνώσεων. Υπάρχει ένα ε, κεφάλαιο που αφορά τις γυναίκες στην Ήπεθρο. Και σε ό,τι αφορά τα αρπακτικά, θέλω να αποζημιώνουμε τους γεωργούς για επιθέσεις ε, από θηρευτές. Δεν θα πρέπει να ε, αγνοούμε αυτό το πρόβλημα και προτείνω αυτή τη λύση της αποζημίωσης. Ξέρω ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, ενισχύσει για το θέμα αυτό, αλλά όχι όλα. Γι' αυτό και προτείνω μια γενική λύση. Να αποζημιώνονται οι γεωργοί που τα κοπάδια τους πλήττονται από επιθέσεις θηρευτών. Επίσης, ό,τι αφορά τα σχέδια. Σε ό,τι αφορά τη δομή και την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων, υπάρχει δυνατότητα να οριστούν περιφερειακές αρχές διαχείρισης για τις παρεμβάσεις της αγροτικής ανάπτυξης και να ληφθεί υπόψη η συνταγματική πραγματικότητα των κρατών μελών. Δηλαδή αυτά τα περιφερειακά σχέδια να συμπεριληφθούν στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Επίσης, διαγράφω την πρόταση για πρημοδότηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ουσιαστικά είναι μια νέα κύρωση που προστίθεται στις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση μη τήρησης των περιβαλλοντικών στόχων των κρατών μελών. Επίσης, ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που συμπεριλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια. Ε, προτείνω εφαρμοστικές πράξεις για τους ε, δείκτες ε, και τους κανόνες εισοδήματος. Προτείνω να είναι καταξιδότηση πράξης και όχι εκτελεστικές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικά στοιχεία στο νέο σύστημα, γι' αυτό και καλό θα είναι να, είναι, υπόκεινται σε καταξιδότηση πράξης. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για την έγκριση των σχεδίων, εγώ διαγράφω τον, κανονισμό, τον μηχανισμό Stop the Clock που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με το ρολόι για να είναι πιο ελαστική η διαδικασία. Αυτό είναι σε γενικέ γραμμέ ε, το έγγραφο που σα πρότεινα. 450 περίπου τροπολογίε έχουν κατατεθεί και περιμένω τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ. Καλώ να περάσουμε στη συζήτηση. Πρώτα θα μιλήσουν οι σκιώδει ηγητέ για δυόμιση λεπτά ο καθένας. Κυρία Νόιχλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια έκανε πραγματικά τεράστια προσπάθεια, έγραψε τροπολογίες, μας παρουσίασε σήμερα ότι το θέμα αυτό πρέπει να το δούμε από πολλές οπτικές. Σωστό είναι αυτό. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν έχουμε βέβαια πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να δούμε ε, τα βασικά σημεία. Τα βασικά ουσιώδη σημεία πρέπει να είναι ε, στον πυρήνα τη συζήτησή μα. Νομίζω ότι ε, το καθήκον μια εισηγήτρια είναι να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, να δώσει ένα μπούσουλα. Και εδώ θεωρώ ότι σε πολλά σημεία έχω αντίθετη άποψη. Είπατε ότι από τη μια ε, θέλετε να υπάρξει κοινή γεωργική πολιτική και πρέπει να μπει στο κέντρο. Απ' την άλλη όμως σε πολλά σημεία μιλήσατε για τις, απο, για τις ε, αποσυνδεδεμένες πληρώμες, ε, για την κατάσταση της ερεσιμότητας Εκεί παραμένετε πάλι σε ένα ασαφές πλαίσιο και μιλάτε για το ότι θα μπορούσε να το κάνει κανείς και θα, ή θα μπορούσε να μην το κάνει. Η κοινή γεωργική πολιτική όμως χρειάζεται ένα πράγμα Καταρχά χρειάζεται μια, ένα συγκεκριμένο όριο για όλα τα κράτη-μέλη. Ανώτατο, το χρεωτικό, τελεία και παύλα. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την ευρωπαϊκή πολιτική και την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Η δεσμευτική αυτή, τα δεσμευτικά αυτά ανώτατα όρια που θα είναι και υποχρεωτικά θεωρώ ότι είναι ουσιώδου σημασία και εσεί στη δική σα την παρουσίαση δεν το βλέπετε έτσι. Θέλετε να υπάρχει ένα εθελοντικό σύστημα. Και από 100.000 και πάνω, λέτε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η άγουσα θα κατακαιρματίσει την κοινή γεωργική πολιτική. Παρόμοιο για τις, για τις ε, για τα περιβάλλον. Πρέπει να είναι υποχρεωτικές για όλα τα κράτη-μέλη, για όλα τα κράτη-μέλη. Υποχρεωτικές. Αν ε, είναι θελοντικές για κάποιους, υποχρεωτικές για κάποιους, τότε δεν θα έχουμε κοινή γεωργική πολιτική η Κομισιόν στους στόχους ε, έχει υποβάλει ε, μια πρόταση που είναι λίγο ασαφής, λίγο φλού. Πρέπει όμως εμείς να έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Εφόσον τους έχουμε, όλες αυτές ή, ε, όλα αυτά τα θέματα για το περιβάλλον θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσω να κάνω μια συνολική αποτίμηση. Η Κομισιόν έχει υποβάλει μια πρόταση και βλέπω ότι αυτή η πρόταση μέσω της εισηγήτριας δεν γίνεται ακόμη πιο ε, ακριβής. Και το, το ερώτημα είναι θέλουμε, είναι ο στόχος μας να έχουμε μια βελτιωμένη πρόταση ή δεν θέλουμε να κάνουμε πιο ακριβή θέματα που μας απασχολούν έτσι ώστε να είναι λίγο πιο σαφή. Συγκεκριμένα, 70% των κορδιλίων για την βιωσιμότητα είπατε, ε, αυτές, αυτό είναι από τις παλιές ε, άμεσες πληρωμές. 70%. Αυτές δεν είναι οι άμεσες πληρωμές όμως που ε, πραγματικά πλήττονται από τον πληθυσμό, από τους πολίτες, που δεν καταλαβαίνει πια γιατί δίνουμε λεφτά ανα ε, επιφάνεια. Αυτές οι άμεσες ε, πληρωμές λέτε ότι θα παραμείνουν στο 70% και θα δίνονται τα κονδύλια ανά επιφάνεια. Ε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούμε, να το ξανασυζητήσουμε. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια ένα κοινό, μια κοινή πολιτική με συγκεκριμένε προποθέσει για την αιρεσιμότητα. Πρέπει να την υποστηρίξουμε. Χρειαζόμαστε οικολογικά προγράμματα υποχρεωτικά και χρειαζόμαστε και αλλαγή των στόχων της κοινή γεωργικής πολιτικής σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική, η οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Ευχαριστώ. Μα ήδη έχουν ε, συναντηθεί οι σκιώδεις ηγητές με την εισηγήτρια και είχαν ε, δυνατότητα να κοινοποιήσουν τα σχόλιά τους ε, στην εισηγήτρια. Ο κύριος Χαϊταμα. Yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια για την ε, έκθεσή της. Κατέβαλε σημαντική προσπάθεια, πολλές τροπολογίες. Ένα-δύο πράγματα τώρα με τα οποία συμφωνώ. Αυτό που λέει για τους εξερχομένους, για την κάλυψη των γυναικών στη Γεωργία, αλλά χρειάζεται να βελτιώσουμε το κείμενο ούτως ώστε να προσανατολίζεται προς τις επιδόσεις, προς τους στόχους η Γεωργία, να συνδεθεί περισσότερο το θέμα των στόχων με τις ε, επιδόσεις και τι θα μας πει το ελεγκτικό συνέδριο ότι δεν, δεν, δεν, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε για τους ε, στόχους μας. Για να συζητήσουμε πρώτα πρώτα το βασικό στόχο της ΚΑΠ που είναι το να μπορούμε να πετύχουμε την ανταγωνιστικότητα για αυτόν τον τομέα και δεύτερον ότι θα πρέπει να προσφέρουμε κοινοφιλή υπηρεσία Έχουμε όλα αυτά, αλλά κολλάμε εμείς ως βασικό μέσο, έχουμε κι άλλα, την ε, ενίσχυση με τις άμεσες πληρωμές. Αλλά υπάρχει το, και το θέμα της διαχείρισης του κινδύνου και άλλες μεταβλητές. Άρα θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους σύστημα ενίχνευσης παρακολούθησης για να βλέπουμε πώς θα πάμε την ανταγωνιστικότητα. Ε, αν δεν κάνω λάθος και για το κλίμα, στο άρθρο 87 προβλέπονταν κάτι τέτοιο. Ε, εκεί έχουμε το σύστημα παρακολούθησης των δαπανών να μην ξεχνούμε να κάνουμε το ίδιο εδώ για την από τους βασικούς της στόχους που είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας να ισχύει η διαλογική και εδώ. Για να δω τώρα τι γίνεται με τα δημόσια αγαθά και αυτό είναι στόχος της γεωργίας, περιβάλλον, κλίμα, ε, βιοπικιλότητα, ύπεθρο στο τοπίο ε, και εδώ ισχύει η αιρεσιμότητα τα οικολογικά προγράμματα, ο δεύτερος πυλώνας. Μα γιατί δεν προσπαθούμε να έχουμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση, γιατί και πάλι επικεντρωνόμαστε στην αιρεσιμότητα και έχουμε και την ε, ενισχυμένη αιρεσιμότητα. Μα εάν κάτι δεν αποδίδει, γιατί να επιμένουμε σε αυτό. Αν κανείς ε, είναι γεωργός και είναι στην ΚΑΠ, ε, θα πρέπει απλώς να τσεκάρει κάποια κουτάκια σε ένα έντυπο για να πάρει από τις Βρυξέλλες τα χρήματα. Για να δούμε όμως. Κολλάμε στις μεθόδους και όχι στα αποτελέσματα. Ε, δεν πετυχαίνει κανείς αποτελέσματα έτσι. Θα πρέπει προσέγγιση να γίνεται με το βλέμμα στον σκοπό, να ωφελείται ο Γιώργος, να του δίνει κανείς κίνητρα να προσπαθεί για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Εγώ αυτό σας προτείνω, να κατεβάσουμε τον πύχη όσον αφορά την αιρεσιμότητα. Να έχουμε οικολογικές στρατηγικές. Να, να κάτσουμε να τα πιούμε και να τα βρούμε με τους πράσινους, γιατί έτσι θα πάμε καλύτερα στα μέτωπα κλίματος, βιοποικιλότητας και αυτά. Α, το είπε ε, η κυρία Νόχλ, νομίζω. Να δούμε τι θα γίνει με τις ενισχύσεις που συνδέονται με τις εκτάσεις με, με, τη γη. Εγώ δεν θέλω αυτό. Θέλω οι καταβολές, οι ενισχύσεις να συνδέονται με τις πράξεις, με τις δράσεις. Ο Πρόεδρος. Ε, ωραία η θεωρία και εύκολο να το πούμε, αλλά δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Πόσο ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Ρασία για την έκθεση. Όταν ήρθα εγώ στην Επιτροπή θεωρούσα ότι θα βλέπαμε ότι αυτοί που θα έπρεπε να πάρουν αυτά τα χρήματα όντως θα τα πάρουν και οι άνθρωποι ας πούμε όπως η Βασίλισσα δεν θα τα έπαιρναν. Εν τω μεταξύ ωστόσο μου έδωσε κάποιες ελπίδες η Επιτροπή και εξεπλάγει από τις απόψεις διαφόρων συναδέλφων. Μάλιστα εξεπλάγει από τις απόψεις και του ΕΛΚ, γιατί μιλούν για προστασία της οικογενειακής εκμετάλλευσης, μιλούμε για το τι απειρημώνεται η Ήπεθρος, μιλούμε για την Επιτροπή Ελέγχου που λένε ότι πρέπει να, είναι καλύτερη, να υπάρχει καλύτερη κατανομή της, ε, της ΚΑΠ, ε, ότι δεν θα πρέπει να ε, μοιράζονται με τους γείτονε τους τα κονδύλια. Δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά όμως εδώ. Στην αρχική πρόταση και τις σε σχέση με τα όσα προτείνει η κυρία Γκαρσία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει είναι το εργασιακό κόστος για το κάπινγκ, για τα ανώτατα όρια. Αυτό θα πρέπει να το απορρίψουμε. Έχουμε ένα σύστημα όπου οι γεωργοί πληρώνονται με βάση του τι, κάνουνε, ε, τι κάνανε πριν από 25 χρόνια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την ανομαλία, γιατί αλλιώ δεν θα υπάρχει τίποτα να ανακατανύμουμε σε αυτού που όντω το αξίζουν και να επιτύχουμε στόχου που είναι πιο επίγοντε. Άκουσα και το ΕΛΚ να λέει τα τελευταία χρόνια. Ε, εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει αυτό όμω γιατί προφανώς δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να διαγραφεί η πρόταση που λαμβάνει υπόψη το εργασιακό κόστος. Επίσης, η αλλαγή στην πρόταση λέει ότι οι βασικές πληρωμές θα είναι 75% του εθνικού μεσουόρου και περνάμε σαν 100% τώρα του, 100, του ναι, μεσουόρου μέχρι το 2027. Στα, οικονομικά, στα οικολογικά προγράμματα, συγγνώμη, είναι, είναι, δεν είναι στοχευμένα, δεν είναι μετρήσιμα, είναι ασαφή και δεν μπορούν να επιδείξουν αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν δράσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα για να μπορέσουμε να τα συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Και γενικώ, ούτω ή άλλω, ο προπολογισμό απειλείται για την αρεσιμότητα που, την, που αντικαταστά, συγγνώμη, αντικαταστά την, την ε, οριζόντια συμμόρφωση. Συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Χόιχελμαν. Μιλούμε για το ότι μετακινούμεθα σε ένα σύστημα, αν δείτε το Gaia 2, για να πάρει κανείς τη βασική πληρωμή, θα πρέπει να, ε, ε, κάνει προστασία, να προστατεύσει τους οικοτόπους ε, κτλ. Άρα δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό. Αυτό θα πρέπει να είναι ειδικό ε, περιβαλλοντικό ε, πρόγραμμα όπου θα πληρώνονται έξτρα μάλιστα αυτοί που το κάνουν. Εγώ προς το παρόν ε, θερμαίνω με συγκεκριμένου τρόπου στο ε, σπίτι μου και ξέρω ότι η κόρη μου που είναι 4 χρονών αυτή τη στιγμή κάθεται μπροστά στο τζάκι και ζεσταίνεται. Αν θέλετε τώρα να δημιουργούμε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορούμε πια να ανάψουμε το τζάκι και δεν θα παίρνει κανένα τίποτα ως αντιστάθμισμα για κάτι που άλλαξε, τότε δεν πρόκειται να αλλάξει το σύστημα. Αυτή η αιρεσιμότητα πρέπει να αλλάξει. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα όπου θα δίνεται κίνητρα, θα δίνει κίνητρα στους ε, γεωργούς. Ε, έχω κι άλλα πολλά να πω, αλλά δεν έχουμε χρόνο, οπότε θα τα βάλω σε τροπολογίες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να εξηγήσω κάτι. Ο κύριος Ντάς δεν έχει ακόμη πάρει το λόγο. Ε, μιλήσατε για κάτι που είχε πει κάποια στιγμή ο κύριος Ντές, αλλά ο κύριος Ντές δεν έχει καν μιλήσει. Ε, χωρίς μικρόφωνο, ο κύριος Φλάναγκαν. Ε, ευχαριστώ, πρόεδρε. Είμαι λίγο απογοητευμένος με τις προτάσεις της ε, εισηγητρίας. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι προσεκτικός. Αδύναμη η πρόταση της Κομισιόν, τώρα επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί μερικοί ωραίοι τίτλοι έμειναν τελικά. Ωραίοι τίτλοι για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, αλλά που δεν έχουν καμιά ουσία. Δυστυχώ πρέπει να το πω αυτό. Αυτέ οι προτάσει δεν λαμβάνουν υπόψη ξεκάθαρα τι μεγάλε κρίσει που έχουμε, την έλλειψη, την απώλεια βιοπικιλότητα, το κλιματικό πρόβλημα το οποίο το αγνοούμε πλέον εντελώ την πρόταση και έχουμε και εξαφάνιση των μικρών εκμεταλλεύσεων. Δεν βλέπω καθόλου να αναφέρονται όλα αυτά. Αν εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για τις ε, νέες αυτές ε, προτάσεις. Η κυρία Γκαρσία λέει ότι θα είναι στο 70% ε, από τον πρώτο πυλώνα. Ε, εντάξει, αυτό είναι βήμα προς τα πίσω όμως. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην κρίση, καμία αναφορά σε σκόπιμη ανακατανομή κονδυλίων. Συμφωνώ με του σοσιαλιστέ που λένε ναι, ανώτατα όρια, αλλά εντάξει, δεν μπορούσαν να το ρυθμίζουν και τα κρατημέλη. Α, δούμε πώ θα γίνει. Ε, δεν θα γίνει καμία, δεν θα τεθούν καθόλου ανώτατα όρια, άμα τα αφήσουμε έτσι φλού. Γι' αυτό Επίση, αν δεν κάνουμε δεσμευτικού του ε, περιβαλλοντικού ε, στόχου και τα αφήσουμε στα χέρια των κρατών μελών για να αποφασίσουν τι είναι σημαντικό και τι όχι, ε, θα, αρχίσουμε να, θα αρχίσουν να μειώνονται όλο και περισσότεροι στόχοι και στο τέλο δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτό φοβούμαι εγώ. Και δεν έχουμε και καμία απάντηση να δώσουμε σε αυτό. Με την κλιματική αλλαγή, τι γίνεται αν δεν θέσουμε δεσμευτικού στόχου για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, για να μειώσουμε α πούμε τι εκπομπέ αερίων. Τι γίνεται με τη βιοπικιλότητα όταν δεν έχουμε υποχρεωτικά μέτρα πρασινίσματο. Και αγνοούνται επίση πληρώ και οι εκθέσει του ελεκτικού συνεδρίου που ακριβώ για αυτέ τι άμεσε πληρωμέ αρχίζει να ε, αμφισβητεί. Μπορούμε να βάλουμε έναν ωραίο τίτλο στο κείμενο. «Αγαπητή Γεωργοί, αγαπητή αγαπητά κρατημέλη, θα πάρετε λεφτά από τι Βρυξέλλε. και κατά τα λοιπά, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν είναι απάντηση όμω αυτό στα θέματα του μέλλοντος, ούτε καν απάντηση για του ε, φορολογουμένου δεν είναι. Για το ποιου στόχου θέλουμε να πετύχουμε. Για, τον, ε, για τους στόχους είπατε ότι ναι, ακόμη κι αν οι στόχοι των κρατών μελών είναι, είναι, είναι κακοί ή δεν επιδευθούν, πάλι δεν υπάρχουν οι κυρώσει. Ε, λοιπόν, γιατί να βάλουν στόχου στα κρατημέλη δεν πρόκειται να τιμωρηθούν σε εισαγωγικά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στόχου που να πρέπει να τηρούνται και να ε, συνοδεύονται και από κυρώσει. Πρέπει να έχουμε κίνητρα όταν προβλέπουμε ε, στόχους. Και αν δεν τους πλήρει ε, κανένας, τότε πρέπει όντως να τιμωρείται σε εισαγωγικά. Αυτό εμένα με εκνευρίζει γιατί πραγματικά δεν ε, βλέπω καθόλου να αναφέρονται. Είχαμε μία ε, μείωση 30%. Έγινε αποδεκτή και τώρα πάει ακόμη πιο πίσω η παραχωρία ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη υπαίθρου. Ε, όλες αυτές οι θετικές προσεγγίσεις που είχαμε δεν αναφέρονται πουθενά και μάλιστα ε, υποτιμώνται κιόλας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν εγώ θα υποβάλω αρκετέ τροπολογίε, αλλά ουσιαστικά πάνε προς την τελείω αντίθετη κατεύθυνση από αυτέ τι ε, συγκέντρες. Ευχαριστώ. Κατά τη γνώμη μου, η θέση της Επιτρόπου, του Επιτρόπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι α, ε, υπέρ των ανώτατων κονδυλίων, των ανώτατων κατοφλίων. όχι την ομοιομορφοποίησή τους, γιατί είναι άλλη κατάσταση στο βορρά και άλλη στο νότο, αλλά δεν νομίζω ότι απάδει πολύ από τη δική μας πρόταση η θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα άνατα τα όρια. Ο κύριος Κάρας κάλεσε εκπροσώπους ε, γεωργών από την Αυστρία, τους καλωσορίζω θερμά στην εδρίασή μας και δίνω το λόγο στον κύριο Τσούλο. Ο κύριος Ταραμπέλα ξεκίνησε τα χειροκροτήματα. Τσούλο, ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την ε, εισηγήτρια. Πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Θα προσπαθήσω να σας τα πω περιληπτικά και να αναδείξω κάποια θέματα για μας πάρα πολύ σημαντικά για αυτή τη μεταρρύθμιση. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να δούμε τι θα γίνει με το εθνικό πρόγραμμα για ούτως ώστε κάθε χώρα να έχει εγγυήσεις ότι κάθε φορά θα γίνεται σεβαστό το τι ενδιαφέρει την κάθε περιοχή. Θα πρέπει επίσης να είναι οι διατάξεις ε, σαφείς, απλές και να υπάρξει μεταξύ κράτους και περιφερειών επικοδομητικός διάλογος και έτσι εγκαίρως να εφαρμοστούν όλα αυτά. Θα πρέπει κάτι να γίνει με τον ορισμό του Γεωργού, να μην είναι ασαφία βέβαια τα πράγματα, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί εδώ το θέμα. Να δούμε τι θα γίνει με αυτούς, οπόμενο πώς θα καλυφθούν αυτοί που σήμερα θεωρούνται Γεωργοί. Επίσης, να δούμε τι γίνεται με τον ενεργό Γεωργό, αυτή την έννοια που υπάρχει στον οριζόντιο κανονισμό. Τώρα όσον αφορά την, ε, τις μεταβολές στη, στα ποσά των πληρωμών να είμαστε μέσα στο πνεύμα το οικονομικό των ημερών θα πρέπει αυτό να το σκεφτούμε καλά. Θα δούμε τι θα γίνει με την εξωτερική σύγκληση. Να μην ξεχνούμε κάποια στοιχεία όπως την διαφορά του κόστους εργασίας από το ένα κράτος στο άλλο και η εσωτερική σύγκληση επίσης θα πρέπει να ενεργήσει να τη χρησιμοποιήσουμε διορθωτικά για κάποιους ιστορικούς τίτλους. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο ανώτατο κατόφλι, είναι σωστή αυτή η προσέγγιση για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Αλλά να μην συνδέονται αυτά τα κατόφλια με την οικονομική συγκυρία, αλλά με τα εθνικά χαρακτηριστικά. Γιατί αυτά διαφέρουν πολύ από το ένα κράτος στο άλλο, το ένα εθνικό σύστημα στο άλλο. Έτσι θα εξασφαλίσουμε με αυτά τα ανώτατα όρια την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Θα δούμε επίσης τι θα γίνει με τις ενώσεις των γεωργών αλλά να μην γίνει αυτό με τρόπο αντιπαραγωγικό. Επίσης, πρόκειται για κοινή πολιτική και αυτό αφορά και τους ελέγχους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών σχεδίων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πλαισίωση των κρατών μελών από την Κομισιόν και έτσι τα εθνικά προγράμματα και σχέδια να κατατείνουν στην επίτευξη των στόχων. Άρα η Κομισιόν, η Ένωση να μην είναι απλώς ο χωροφύλακας, αλλά να βοηθά αυτή την κοινή προσπάθεια. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε το γύρο των σχεδόν εισηγητών. Τρία λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μίλησε κατά μέσο όρο κάθε σκιώδη εισηγητής. Περάμε στους λοιπούς ε, ευρωβουλευτές, 1,5 λεπτό ο καθένας. Ο, ο κύριος Κολομπιέ. Ή δεν θέλετε το λόγο. Όχι, οπότε ο κύριος Ντές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τη συνάδελφο για την παρουσίαση της έκθεσης. Σε αντίθεση με την πρόταση της Κομισιόν, εδώ υπάρχουν πολλές βελτιώσεις μέσω τροπολογιών. Θα φροντίσουμε να υπάρξουν κι άλλες να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η πρόταση. Ένα σημείο θα ήθελα να σχολιάσω για την ε, πρόθεση και την ενίσχυση των νέων γεωργών. Θα θέλαμε εδώ μέσω του δεύτερου πυλώνα να κάνουμε μια καλύτερη επένδυση ή πρόθεση των ε, ε, επενδύσεων. Μπορεί μια εκμετέλεύση να είναι πιο καλά οργανωμένη και να μπορεί να τύχει καλύτερης επένδυσης Υπάρχει μια άλλη εκμετάλλευση που ε, χρειάζεται όμως την επένδυση, αλλά δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα για να την αποκτήσει. Α, ε, μπορεί λοιπόν η μία εκμετάλλευση να χρειάζεται πιο άμεσα την ε, επένδυση. Θα πρέπει να δούμε και το, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα κάνουμε τις επενδύσεις. Η Κομισιόν λέει ότι τιμωρούνται οι χώρες οι οποίες μέχρι τώρα ε, μέσω του δεύτερου, πυλώνα ε, έπαιρναν πολλά χρήματα για τα, από την ε, από την ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, ας πούμε το Νότιο Τυρόλο ή στην Γερμανία ε, κρατήδια. Πλέον δεν θα μπορούν να δίδονται πληχιά αυτά τα κονδύλια για ας πούμε τετραετή, πενταετή προγράμματα. Αν αυτό είναι υποχρεωτικό, τότε σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον κονδύλια από τον δεύτερο πυλώνα. Επίσης, για την αρμοδιότητα των κρατών μελών και τα περιβαλλοντικά προγράμματα. Εδώ ε, νομίζω ότι ουσιαστικά μετακυλίουμε την ε, γραφειοκρατία από την Ευρώπη πάει στα κρατη Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι αυτό. Αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Αυτό το μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Αν παραμείνει έτσι, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω. Πρέπει να αλλάξουν πολλά ω προ αυτό, έτσι ώστε η πρόταση αυτή να μπορεί να τύχει τη στήριξή μα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί αλλιώ δεν θα μου μείνει τίποτα άλλο, αλλά να καταψηφίσω το σύνολο της πρότασης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα, να ευχαριστήσω την κυρία Εράνθη, γιατί ήταν ε, μνημειώδες αυτό το οποίο έκανε πάνω από 400 τροπολογίες, ε, βέβαια, και μας αρέσει το ότι θέλει να πάμε μέχρι το 2023 με αυτήν την ΚΑΠ. Ανάγκη αυτό, δεν είναι δυνατόν κάθε δύο χρόνια να τα αλλάζουμε όλα. Πάντως ε, σε αυτό το λεπτάκι που έχω θέλω να σας πω ότι ακόμα νιώθω κάποια μηχανία, μια απορία, όχι τόσο στην ουσία, αλλά το πρόβλημά μου είναι η θεσμική αρχιτεκτονική αυτής της μεταρρύθμισης. Συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε με αυτά τα στρατηγικά σχέδια να αποκτήσουν αρμοδιότητες στα κράτη όσον αφορά τη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ. Επανεθνικοποίηση. Θα είναι αυτό όμως απλούστευση. Λέμε ότι έχει γίνει απλούστευση εδώ στις Βρυξέλλες. Πούντι, δεν τη βλέπω. Αυτό και τους ε, Γιώργους. Λέμε ότι θα έχουμε ε, μια διαχείριση για πρώτο και δεύτερο πυλώνα ε, όμως τριμώχονται στα κρατημέλη, ε, προβλέπουν στο συνταγμά τους κάποια κρατημέλη, ε, των τούτων στις περιφέρειες και επομένως πριν μπούμε στο λαβύρινθο αυτής της μεταρρύθμισης να δούμε αν είναι αυτό που θέλουμε η πανεθνικοποίηση. Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Γιατί ο ρόλος μας αυτός είναι, η ΚΑΠ. Και βλέπουμε ότι τώρα η διαχείριση θα γίνεται από κράτος μέλος και κομισιόν. Δεν είναι αυτή η πρόταση Ντόσμαν. Θα πρέπει το πρώτο που έχουμε να κάνουμε πριν μπούμε στην ουσία να ξεχαδέσουμε αυτό που σας λέω και μετά να δούμε ποιος είναι ο ρόλος μας. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω το έργο της συγκεκριάς μας. Γιατί ε, μέρημνα της είναι να πλουστεύσει τη ζωή των γεωργών και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Νόιχλ, διαφωνώ ριζικά μαζί σας. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε το βιοαβίωτο το στους γεωργούς, αλλά να τους επιτρέψουμε να ζουν εξεπρεπώς ασκώντας το επάγγελμά τους. Οι καταναλωτές ε, είναι όλο και πιο απαιτητικοί στις προδιαγραφές ε, που ζητάνε για το τρόφιμά τους και ταυτόχρονα κάνεις δεν θέλει να πάει στην Ήπεθρο να ασχοληθεί με τη γεωργία γιατί το 1 τρίτο των γεωργών ε, δεν λαμβάνει καν το ελάχιστο μισθό που έχουν τα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να διατρανώσω ότι στόχος μου είναι να επαναφέρουμε την αξιοπρεπία στο γεωργικό επάγγελμα και όχι να ψήσουμε το ψάρι στα χείλη των γεωργών. Επίσης, η γεωργική μας πολιτική θα πρέπει να είναι όντως κοινή γεωργική πολιτική. Και συμφωνώ με τα σχόλια του κ. Ντεκάστρο. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να είναι καλύτερα πλαισιωμένα και να διασφαλίσουν αυτό το κοινό χαρακτήρα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειε. Θα πρέπει σε όλες τις χώρες ε, με τον ίδιο τρόπο να συμπαραστεκόμαστε στους γεωργούς. Και θέλουμε και ένα οικονομικό σκέλος που θα δράζεται και στις άμεσες στραματικές ενισχύσεις, αλλά και όπως είπε και ο, Αλμπερντές, θα πρέπει να έχουμε μια πραγματική πολιτική για να ε, ευνοούμε τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, ήδη έχουμε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και το οικολογικό πρόγραμμα που προτείνεται θα πρέπει ε, να παρακολουθεί γενικώ τις, ε, τις εξελίξεις ε, της φάρμας, τις γεωρικές εκμεταλλεύσεις, αλλά να μην είναι ένας πλέον όρος που υποβάλλεται για τη στρεματική ενίσχυση. Επίσης, θα πρέπει σε ένα παράρτημα να έχουμε τις ψαλίδες των ενισχύσεων που μπορεί να δίνει κάθε χώρα. Ή δεν θα έχουμε για τις ίδιες καλλιέργειες και για τις ίδιες καταστάσεις πολύ διαφορετικές ενισχύσεις. Με αποτέλεσμα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 και το συνάδελφο Ντεκάστρο. Συμφωνώ απολύτω μαζί του και θα ήθελα τέσσερα συγκεκριμένα σημεία να σχολιάσω. Καταρχά. πρέπει να δούμε πώς η Κομισιόν θα εγκρίνει αυτά τα στρατηγικά σχέδια έτσι ώστε οι αρμοδιότητες να ε, να μην υπάρξει κατάχρηση των αρμοδιοτήτων και να υπάρξει καταπίεση των ε, κρατών μελών. Δεύτερον, η ανακατανομή και η, δίκλη, η κλίδα αυτή ανακατανομής. Ε, μιλάμε για ε, εθελοντική σύνδεση, η οποία εξαιρείται πια από τις, ε, από το, από τις διατάξεις. Τρίτον, η, αυτή η, επιδότηση νομίζω ότι ανταγωνίζεται άλλες διατάξεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει τα δύο, από τα δύο συστήματα να μπορούν να επιλέγουν ένα τέταρτο. Προς το παρόν τα κράτη-μέλη θα έχουν ε, πρόβλημα με την, ίδρυψη, λόγω της, ε, με την άρδευση λόγω της ε, κλιματικής αλλαγής. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε ίσως νέες εγκαταστάσεις άρδευσης, ανεξάρτητα βέβαια και από τον όγκο των υδάτων που, υπάρχει, που υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν και εγκαταστάσει εξοικονόμηση υδάτων. Αυτά και ευχαριστώ. Η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με τα σχόλια του κυρίου Ντεκάστρο και του κυρίου Νταντά. Γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θα ήθελα να συγχαρώ και την εισηγήτριά μας, την κυρία Γκαρσία, για την πολύ ενδιαφέρουσα και εργόδη προσπάθειά της. Και συμφωνώ σε πολλά σημεία με την εισηγήτρια. Φυσικά έχω και κάποιες διαφωνίες, κυρίως στην περισσότερη επικορικότητα στα κράτη-μέλη. Ούτε με την πρόταση για το κάπινγκ συμφωνώ, κυρία Ελλάς Γκαρσία. Και το εξήγησε καλά η κυρία Νόιχλ. Εμείς προτιμούμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή το κάπινγκ, τα ανώτατα όρια, να ορίζεται σε κεντρικό επίπεδο Βρυξελών και όχι ε, κάθε χώρα να επιλέγει το ανώτατο όριο που τη βολεύει ξεκινώντα από την αφετηρία των 100.000. Προτιμώ την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κάπινγκ. Θα πρέπει να είμαστε αυστηροί και να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθορισμό των ανατάτων όριων. Συμφωνώ με την πρότασή σα για το ρόλο τη γυναίκα στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην παρουσία των γυναικών στι αγροτικέ ζώνε. Και όχι μόνο για, την, για τον απαραγωγικό του ρόλο, για το ότι είναι μητέρε, αλλά και για το έργο που προσφέρουν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, που αγνοείται πλήρως. Είναι τελείως ε, άδειλος ο ρόλος τους μέχρι στιγμής. Θα καταθέσω λοιπόν σχετική τροπολογία. Επίσης για τους νέους αγρότες δεν βλέπω να είναι νέος κάποιος που είναι 45 χρονών, ούτε παρατείνοντας την ηλικία των ε, αγροτών για τον ορισμό του νέου αγρότη θα φέρουμε περισσότερους αγρότες στην γεωργία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παροτρύνουμε τους νέους ε, και τις ε, νέες ερχόμενους να εισέλθουν. Επίσης για, τις, ε, για τον ενιαίο φορέα διαχείριση θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο ρόλο στις περιφέρειες. Και κάτι που δεν αποσαφηνίστηκε με τις διεκθέσεις. Νομίζω ότι είναι σωστό να λαμβάνουμε υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει η οργάνωση των γεωργών γιατί πραγματικά οι ιδιαιτερότητε των συνεταιρισμών είναι που πλουτίζουν τον κλάδο. Θα πρέπει να φέρουμε χωριστή τροπολογία για το θέμα αυτό. κύριο Καλινόφσκι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητριά μα, γιατί πραγματικά είναι τεράστια προσπάθεια που έκανε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερω την κυρία Γκαρσία που πρότεινε να ε, διατηρηθεί το ανώτατο όριο ε, σε ό,τι αφορά την ε, στήριξη της παραγωγής. Πολύ καλή πρόταση και την υποστηρίζω. Το ίδιο θα πρέπει να εφαρμόσουμε και στην περίπτωση της ελαστικότητας μεταξύ των πυλώνων και η δυνατότητα μεταφοράς 25% ε, είναι καλή και δικαιολογημένη πρόταση και ούτε ε, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οξύνη των τη διαμάχη των, γεωργών. Αυτό που πλήττει τον ανταγωνισμό είναι οι τεράστιε διαφορέ ε, στα επίπεδα άμεσων ε, ενισχύσεων που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ χειρότερο για τον ανταγωνισμό. Σε ό,τι αφορά την ε, υποχρεωτική διάθεση για τα κράτη-μέλη, δηλαδή τα στρατηγικά του σχέδια να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τον ορισμό του γνήσιου αγρότη, δηλαδή του αγρότη που πραγματικά ασχολείται με τη γεωργία. Θα προτιμούσα να έχουμε κεντρικό ορισμό και όχι κάθε χώρα να ορίζει όπως θέλει το γνήσιο Γιώργο, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μεγάλες διαφορές αν υπάρχουν διαφοροποιημένοι ορισμοί. Και γι' αυτό θα καταθέσω και τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συγγετρία για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Ήταν πραγματικά πολύ περίπλοκη η εργασία που χρειάστηκε να κάνει. Αλλά πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Όπως και ο Παύλο, θα ήθελα και εγώ να πω ότι σήμερα θα έπρεπε να μιλούμε για α, τις λεπτομέρειες για το, αυτό την ε, νέα delivery, το νέο delivery model. τώρα Νομίζω ότι έχουμε συζητήσει για όλα τα υπόλοιπα πλην αυτού. Ε, μιλούμε για πιο τεχνικά θέματα, αλλά στη φάση αυτή που είμαστε και που είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε τροπολογίε, νομίζω ότι θα πρέπει να συντονιστούμε λιγάκι καλύτερα μεταξύ των ομάδων για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο αυτό για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα. Θα πρέπει να είναι όντως κοινή η γεωργική πολιτική. Ξέρω ότι ε, συνηθίζω να μακρηγορώ, αλλά θα έπρεπε να μιλήσουμε και για τον ορισμό του γεωργού. Θα πρέπει να ε, είμαστε σίγουροι ότι αυτός που λέει ότι είναι γεωργός το βασίζει σε αντικειμενικά κριτήρια. Πρέπει να δούμε επίσης το θέμα της αρεσιμότητας, πρέπει να το ενισχύσουμε και το θέμα των ενότητων ορίων και της υπαναχώρησης. Ε, συμφωνώ με αυτές τις αρχές, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μη συνδεδεμένες πληρωμές. Και τέλος, για τις συνδεδεμένες πληρωμές, έχουν προταθεί κάποιες τροπολογίες για το άρθρο 30, το οποίο δίνει την επιλογή συνδεδεμένων πληρωμών για έναν ε, μακρύ κατάλογο τομέων, δεδομένου και του νέου delivery model. Αυτές οι εξαιρέσεις εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτες. Ευχαριστώ. Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την εισηγητήρια και έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Καταρχήν, στο στόχο 8 του κειμένου που λέει να προωθήσει την απασχόληση, την ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ε, ανάπτυξη των γεωργικών ε, περιοχών συμπεριλαμβανομένης και της γεωργικής οικονομίας και της δασοκομείας. Λυπάμαι όμως που οι προτάσεις που έγιναν δεν λαμβάνουν υπόψη αυτό το στόχο. Η γεωργία και η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικές φιλοδοξίες και οικονομικές φιλοδοξίες για την δραστηριότητα αυτή. Και πιστεύω ότι η Γεωργία θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στην οικολογική μετάβαση και να μην πω ότι θα πρέπει να είναι και ο κινητήριος μοχλός του περιβαλλοντικού, του οικολογικού μετασχηματισμού. Και δυστυχώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρασε στον ντούκου αυτές τις προτάσεις. Άκουσα τα σχόλια των κυρίων Νταντά, Ντές και Ντεκάστρο και λυπάμαι και εγώ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για τις πρωτεϊνόχες καλλιέργειες γιατί χωρίς τέτοιο σχέδιο θα συνεχίζουμε να εισάγουμε το 70% των φυτικών πρωτεϊνών που μάλιστα θα είναι γενετικώς τροποποιημένες και προέρχονται περισσότερες από, τις, ε, από την Αμερική. Και έτσι δεν θα εξασφαλίσουμε την επιστημιστική μας αυτάρκεια που πραγματικά την αξίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην καλλιέργεια πρωτεϊνών. Ευχαριστώ, δεν θα επεκταθώ άλλο γιατί ξεπέρασα το χρόνο. κυρία Σένορα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Εστέρ για την έκθεσή της. Μια και έχουμε ελάχιστο χρόνο, θα πάω κατευθείαν στο ψάχνο. Από τη συζήτηση μας λείπουν κάποιοι μηχανισμοί προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια τιμή που θα ανταμείβει τους γεωργούς άνδρες και γυναίκες για το έργο τους και δεν θα είναι τιμή κάτω του κόστους. Γιατί τα δημόσια κονδύλια όλο και μειώνονται και τελικά ε, καταλήγουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας, μεταξύ των περιφερειών, των κρατών και μεταξύ των γεωργών για να μοιραστούμε αυτά τα πενιχρά κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα θετική δράση και την ε, επαγγελματική αναγνώριση των γυναικών τη υπαίθρου, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται στην οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση, η αναγνώριση αυτή είναι σημαντική. Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση των νέων και του νέου ερχόμενου στη γεωργία, ανεξάρτητα από την ηλικία, του ενδιαφερόμενου. Είναι σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει να προκαταβάλουμε τις ενισχύσεις για να μπορούν ε, οι άνθρωποι να ασχοληθούν με την ε, εκμετάλλευση αντί να ε, ξοδεύουν χρήματα πληρώνοντας τόκους στις τράπεζες αφού αναγκάζονται να πάρουν δάνεια. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει πραγματικά να γίνει μια ανακατανομή των ενισχύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σημαίνει κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων και προσδιορισμός πολύ πιο χαμηλών ορίων και υποχρεωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θα έλεγα τρία επίπεδα ανωτά των ορίων. Για τις ορεινές περιοχές υψηλότερο, δεύτερον για τις μειονεκτικές περιοχές και τρίτον για τις λοιπέ περιοχές. Τρία διαφορετικά επίπεδα ανωτά των ορίων. Επίσης, πρέπει να συνδέσουμε την πληρωμή των ενισχύσεων με σαφή μοντέλα που θα είναι φιλοπεριβαλλοντικά και θα συμβάλλουν στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Τίποτε πέραν αυτόν τον στόχο θα πρέπει να αξίζει η ενίσχυση. Σε ευχαριστώ, κύριο Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ΕΣΤΕΡΑ έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά, συμπεριέλαβε πολλά ενδιαφέροντα σημεία, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα βασικό πρόβλημα και ε, το είπαν πολλοί συνάδελφοι. Ε, ούτε η Κομισιόν το έλυσε, ούτε η έκθεση της συναδέλφου και οι τροπολογίες. Η κατανομή, το ε, πρώτο πινώνα, τα 40 δις ε, κάθε χρόνο, τα, ε, τα, κατα, τα με βάση ένα κριτήριο το οποίο είναι παλιό και ανεπαρκές, με αυτό της επιφάνειας δηλαδή. Αν έχετε 20 εκτάρια γη, κάπου σε μια ωραία θέση στην Ευρώπη και την έχετε κληρονομήσει από τους γονείς σας και έχετε και κάποια δέντρα ή θάμνους κτλ μπορείτε να ε, την ε, σκάψετε, να την οργώσετε, μπορείτε να φυτέψετε και να πάρετε και πολλά λεφτά για, τις, ε, για τα 20 εκτάρια. Μπορείτε να δημιουργήσετε. μπορεί τώρα κάποιο με 20 εκτάρια να θέλει να φτιάξει μια οικογενειακή επιχείρηση, να δημιουργήσει θέσει εργασία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια εσωτερική σύγκληση ουσιαστικά. Γιατί το πρώτο κομμάτι της α, έκθεσης για την καλή θέση που μπορεί να βρίσκεται η εκμετάλλευσή σας, την, ε, το, του συμπεριφερόμαστε με πολύ, καλύτερη, με πολύ καλύτερο τρόπο από τη δεύτερη περίπτωση του ανθρώπου που θέλει να φτιάξει την οικογενειακή επιχείρηση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το σκεφτούμε. Ή, ή μετά το ε, μεσημεριανό θα πρέπει να συζητήσουμε με το ελεκτικό συνέδριο για αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτό το σύστημα πια δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε πια και στους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος με, την, με, μεγάλες περικοπές στο δεύτερο πυλώνα και είμαι υπέρ ή υγεωργή που θέλουν να αντιμετωπίσουν επιθέσεις από ε, ε, αρπακτικά, ε, αρκούδες, ε, λύκους κλπ. να αποζημιώνονται. Αλλά τώρα από πού θα αποζημιώνονται, ε, θα πρέπει να το, τώρα να πρέπει από μόνος του να πληρώσει τα έξοδα αυτά ο Γιώργος, νομίζω ότι είναι λάθος προσέγγιση. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την ζημία να την καλύπτει, την ίδια τη ζημία να την καλύπτει και ο Γιώργος. Η κυρία Κατάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Τα λέει πολύ ισορροπημένα και είναι σημαντικό να υπάρχει περιθώριο προσαρμογής από πλευράς κρατών μελών γιατί ισχύουν διαφορετικά σε κάθε κράτος μέλος. Στο στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να μπορούν να διαφοροποιηθούν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να ξυγχρονίσουμε. Βεβαίω και είναι πολύ σημαντική τη σήμερα μέρα η επικουρικότητα και λέμε τώρα για το ποιο θα είναι ο ορισμό του αυθεντικού, του πραγματικού Γεωργού και συμφωνώ με την εισηγήτρια να συνεχίσει να ισχύει αυτή η ενίσχυση που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και φυσικά να ισχύουν τόσο προβλέπει ο ΠΟΕ. Τώρα να... υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά ε, την περίοδο προσαρμογή στη μεταβατική περίοδο που λέμε ότι θα πρέπει να μετατεθεί στο μέλλον και για τις δράσεις για το κλίμα, για το περιβάλλον, ε, ότι θα πρέπει να αποστείλουν το δεύτερο πυλώνα, να μην έχουμε επίσης ε, την απορρόφηση των υπογείων υδάτων όπως προβλέπεται τώρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη ακριβώς τις οι δύο μορφίες της γεωργικής παράδοσης να μην γίνει περικοπή των ενισχύσεων που συνδέονται με την παραγωγή να μπορέσουμε ε, εάν κάποιοι θέλουν να έχουμε προαιρετικές όχι αναγκαστικές ρυθμίσεις όχι ε, ε, κάνουν πολύ περισσότερα οι γεωργοί από το να συμπληρώνουν τις αιτήσει για τις επιδοτήσεις προστατεύουν το περιβάλλον και πολλά άλλα οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη ε, να προτάξουν τις ιδιορυθμίες τους και αυτές να ληφθούν υπόψη. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Γιατί είπατε ότι οι γεωργοί μπορούν να κάνουν περισσότερα από αυτά που περιμένει από αυτούς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σας δώσουμε την ευκαιρία να το κάνουν. Κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ. Για την πανεθνικοποίηση ήθελα να μιλήσω, που την επέκρινε η αλλά βέβαια αυτό δεν αρκεί στο ένα ή στο άλλο σημείο να γράψουμε κάποια πράγματα, θα πρέπει να πάμε στα άρθρα, θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρεια και να έχουμε ελάχιστα πρότυπα τα οποία για, όλους τους, ε, όλα τα κράτη θα ισχύουν εξίσου. Για την καλύτερη βιοποικιλότητα, για, καλύτερο, για καθαρότερο αέρα, για καθαρότερα νερά. Θα πρέπει να δούμε δείκτες, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ναι, θα μετρήσουμε αυτές τις ε, επιχειρήσεις που πήραν μέρος στο πρόγραμμα. Όχι, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένους στόχους. Όπως ας πούμε στο παράρτημα 1 που είναι γενικόλογο. Θα πρέπει να πούμε πόσα, τι ποσοστό θέλουμε, τι μείωση θέλουμε να πετύχουμε για τα αέρια του θερμοκηπίου, ας πούμε. Πρέπει να καθορίσουμε πόσα λεφτά θέλουμε να δώσουμε για το κλίμα, πόσα λεφτά θέλουμε να δώσουμε για την α, α, μείωση προς τα κάτω. πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε, λέμε, τι εκμεταλλεύσει. Ναι, αλλά αν θέλουμε όντω να τι ε, ε, προστατεύσουμε, θα πρέπει να τι ε, εξοπλίσουμε για το μέλλον. Θα πρέπει να προσαρμοστούν σε, σε αλλαγέ κλιματικέ, περιβαλλοντικέ και κοινωνικέ για το πώ εξελίσσονται οι περιφερειακέ περιοχέ. Αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα. Πρέπει τώρα να αρχίσει η δουλειά αυτή, γιατί μιλούμε για 70% άμεσε πληρωμέ και τα υπόλοιπα περνάνε έτσι στο στο παραλίλω ε, δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε τίποτα. Θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πόσα λεφτά για το κλίμα, πόσα για την αναδιάρθρωση, για την ανακατανομή προ τα κάτω, πόσα κονδύλια, άμεσε πληρωμέ. Δεν μπορεί να μείνει στο 70% το ποσοστό αυτό. Γιατί αλλιώ δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Ελάχιστα πρότυπα λοιπόν και συγκεκριμένα ποσοστά κονδύλια για να ξέρουμε τι γίνεται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σε σχέση με τα όσα είπε η συγκήτρια, ε, για ένα σημείο διαφωνώ. Έχουμε φτηνά τρόφιμα σήμερα. 10% ε, φεύγει από τον προπολογισμό μας ε, ή από τα εισοδήματά μας για τα τρόφιμα και είπατε να είναι ακόμα πιο φτηνά τα ε, τρόφιμα, δηλαδή ακόμη χειρότερε τιμέ για του γεωργού. Και αυτό σημαίνει καλή, ακόμη χειρότερη αξιολόγηση ε, τη δουλειά που κάνουν. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό ε, για την παραγωγή των τροφίμων ε, από τους γεωργούς. Είναι ο λάθος δρόμος. Η κοινωνική, κοινωνική πολιτική μέσω φτηνών τροφίμων δεν είναι ο τρόπος που θα πρέπει να προωθήσει η Επιτροπή Γεωργίας. <coughs> Θέλουμε καλές τιμές για τους παραγωγούς. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Τώρα για το κάπινγκ, για τα ανώτατα όρια. Δεν, τα, το καταστήσουμε υποχρεωτικά για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Θα έχουμε ανταγωνισμό και στρέβλωση του ανταγωνισμού επίσης αν, το, αν θέλουμε όντω να εφαρμόσουμε το κάπινγκ, θα πρέπει να ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και αν είμαστε σοβαροί με αυτά που προτείνουμε για τι μικρομεσαίε εκμεταλλεύσει, θα πρέπει να τι υποστηρίξουμε και ποιο τελικά ε, όντω ε, υποστηρίζει το κάπινγκ ή όχι. Θα πρέπει να εμείνουμε στο στόχο μα. Το 70% για την ε, ενίσχυση των εκταρίων, το είπε και ο κ. Ντόρφμαν, είναι μια πολιτική που δεν επιτυχάνει αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. για τις, ε, περιοχές, για τις εκμεταλλεύσεις της περιοχές και ουσιαστικά ε, θέλει φτηνά, φτηνές πρωτεσίλες για τη βιομηχανία. Αν επιτρέψουμε αυτές τις μειώσεις για τη γεωργία, τότε βλάπτουμε όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέσω άμεσης θέσης εμπορίας, μέσω ε, των επιχειρήσεων επεξεργασίας και δεν ενισχύουμε την γεωργία. Νομίζω ότι λοιπόν θα υπάρξουν αρκετές τροπολογίες ως προς αυτό από τη δική μας την πλευρά και ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να χαιρετήσω το έργο της κυρίας Συγητρίας. Να πάω στο βασικό μου μέλημα, το κάπινγκ, τα ανώτατα όρια. Νομίζω ότι πολλοί ε, αγρότες θα επηρεαστούν από αυτό. Και αν μείνουμε στη λογική της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ηγετρίας, ε, θα γίνουμε μάρτυρες πολλών πτωχεύσεων, γιατί οι Γεωργοί στη Ρουμανία, τις κατοχώρες, στη Γαλλία, έχουν συνάψει δάνεια που δεκαετή πρέπει να τα επιστρέψουν όταν ε, συνήψαν αυτά τα δάνεια έλαβαν, είχαν λάβει υπόψη τη, τα δικαιώματά τους από τις άμεσες ενισχύσεις. Αν μετά το 2020 θα περικοπούν αυτά τα ποσά, θα χρεοκοπήσουν οι γεωργοί δεν θα μπορέσουν να αποπληρώσουν τα δάνειά του. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη στα επίπεδα που θα θεσπίσουμε για τα ανώτατα όρια. Και πιστεύω ότι θα πρέπει τα, τα ανώτατα όρια να θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι κάθε χώρα να θεσπίζει τα δικά τη. Επίση, θέλουμε μια ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι άμεσε ενισχύσει. Γιατί όλοι οι γεωργοί στην ίδια αγορά διαθέτουν τα προϊόντα του. Θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό που να συνδέεται με την παραγωγικότητα, όπως είπε ο κύριος Ντόρφμαν. Δεν αρκεί να λαμβάνεται υπόψη μόνο η έκταση. Επίσης θα πρέπει στη συγκεκριμένη έκταση να παράγονται τρόφιμα που ζητούν οι καταναλωτέ Σε ό,τι αφορά τους ενεργούς αγρότες και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε τα κονδύλια να πηγαίνουν σε ανθρώπου που πραγματικά έχουν γεωργική δραστηριότητα, όχι σε κερδοσκόπου ή σε άτομα άσχετα με τη γεωργία. Σε ό,τι αφορά τους θηρευτές, ας μην ξεχνούμε ότι οι θηρευτές δεν είναι μόνο άλλα άγρια ζώα, αλλά προσοχή σε όσους καταστρέφουν τις γεωργικές καλλιέργειες. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ γραφεία για την έκθεσή της, για αυτά τα στρατηγικά σχέδια Αναδύονται κάποια ερωτηματικά γενικώ, γιατί πρόκειται για αυτή την ε, κοινή διάσταση που συρρυκνώνεται, ε, γιατί πρόκειται για βασικό θέμα της Ένωσης. Και ε, επομένω θα πρέπει να εξετάσουμε αυτή την, την πρόταση ε, της εισηγήτριας Σε αυτή την πρόταση της ε, Επιτροπής, δεν συμφωνώ με αυτή την λογική να αποσυνδέσουμε τις κοινέ διατάξεις από τα τα ταμεία. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, άρα θα πρέπει η πολυρύθμιση να επανέλθει η Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις ε, περικοπές του δευτέρου πυλώνα για την ανάπτυξη της υπαίθρου και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με, την, με τον περιορισμό μεταφοράς πόρων τον τρίτο στον πρώτο πυλώνα ε, εγκυμονεί κινδύνου για τον δεύτερο πυλώνα άρα θα πρέπει στο 5% να μείνουμε όσον αφορά τη μεταφορά από τον δεύτερο στον πρώτο. Είναι πολύ σημαντικό τώρα όσον αφορά το οικολογικό πρόγραμμα, τη στρατηγική, την πολιτική θα πρέπει να δούμε αν αυτό είναι κίνητρο για τους γεωργούς, και στη συγχρηματοδότηση να έχουν το δικό τους κομμάτι τα κράτη-μέλη ε, αλλά όχι στο δεύτερο πυλώνα που είναι σημαντικό αυτό. Επίσης για τα πρωτεϊνούχες καλλιέργειες έχει προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν αυτό είναι η σωστή κατεύθυνση και θα δούμε τι θα γίνει με τις συνδυόμενες ενισχύσεις ανατομέα αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί και άρα να προσέξουμε ε, τον τομέα αυτών γιατί έχει στρατηγική σημασία όπως οι προλαλήσαντες συνάδελφοι τόνισαν. Ευχαριστώ. Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσα περισσότερα ακούω τόσο πιο δύσκολο φαίνονται τα πράγματα. Άμα αποσυνδέσουμε τις πληρώσεις από την παραγωγή πρέπει να δούμε με τι προϋποθέσεις θα συνδέσουμε τις πληρωμές στην έκταση στη γη. Θέλουμε να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτούς που έχουν ως πλήρη απασχόληση τη γεωργία. Την τελευταία φορά είχαμε σύγκληση, είναι θέμα εισόδηματός τους. Α, οι κτηνοτρόφοι που παράγουν βόλιο, κρέας και έχουν εγωπρόβατα, έχουν 72 100% του εισοδήματός τους από τις άμεσες πληρωμές. Άρα, ό,τι περικοπεί από εκεί θα είναι περικοπή στο εισόδημά τους. Έχουμε μια τροπολογία για τον ορισμό του πραγματικού Γιώργου. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι δομές θέλουν στη γεωργία τους τι θα κάνουμε με αυτούς που έχουν πλήρη απασχόληση τη γεωργία. Επίσης να μην γίνεται οι κύριοι του ακινήτου να λαμβάνουν την ενίσχυση και όχι η γεωργοί. Να μην γίνεται στην τελευταία μεταρρύθμιση. Τώρα όσον αφορά το περιβάλλον έχουμε την ερεσιμότητα, το πρόγραμμα για το περιβάλλον, αλλά ξέρετε, όταν ο Θεός έπρεπε τον κόσμο, δεν τον χώρισε σε τρία διαφορετικά κομμάτια. Άρα να κάτσουμε να σκεφτούμε τι λέμε στους γεωργούς. Γιατί όταν ε, τους λέμε τι θέλουν να κάνουν για το περιβάλλον, αυτά που τους λέω δεν τα καταλαβαίνουν. Ο κύριος Άγνιο. Ευχαριστώ. Την τελευταία τετραετία εδώ στην Επιτροπή ποτέ δεν είδα με τόση ζέση να θέλουν οι συνάδελφοι να υπαγάγουν την δασοκομεία στην ε, Ιουρία. Μα δεν είναι αρμοδιότητα ε, κοινοτική. Ποτέ δεν συμφώνησε η Επιτροπή μαζί μου. Αλλά τώρα φτάνουμε στο κέριο σημείο που να έρχεται η Επιτροπή και μας λέει συμπαθάτε με δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε τη δασοκομεία. Αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν στο Συμβούλιο να αλλάξει η συνθήκη και αυτό ομόφωνα. Εμέγα να γίνει αυτό να σταματήσουμε να συζητάμε για την δασοκομεία τώρα, για τα πρωτεϊνούχα. Ναι, όντως υπάρχει έλλειμμα και τα περισσότερα από αυτά τα είναι τα όσπρια ε, και είναι συνήθως παραπροϊόντα του βασικού ε, φυτού. Ε, υπάρχει ε, εκπομπή αζότου οξυδίου του αζώτου τέλο πάντων και τους λέμε από τη μία μεριά ε, ε, ότι επισύρει και οι Ρώσοι το να μην μειώσουν τις εκπομπές, από την άλλη λέμε ότι πρέπει να αυξήσουν τα όσπρια και θέλουμε να τους δώσουμε και πηδώματα γι' αυτό. Δηλαδή ό,τι τους δίνουμε το ένα χέρι το παίρνουμε με το άλλο. Δεν είναι αντίφαση αυτό. Ας κάνει κάποιο κάτι επιτέλους γι' αυτό. Ο κύριος Ανδρία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, αρκετοί στην Επιτροπή μας αντιταχθήκαμε από την αρχή στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί κατά τη γνώμη μας δεν ανταποκρίνεται στο στόχο της διασφάλισης του γεωργικού εισοδήματο. ούτε με τις αποσυνδεδεμένες ή τις τρεματικές ενισχύσεις θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε παρκές γεωργικό εισόδημα. Και ταυτόχρονα έχουμε επιστηστικές προκλήσεις περιβαλλοντικές, ανθρώπινες υγείας και ούτω καθεξής. Πάντως, χαίρο την εισηγήτρια γιατί μπήκε στις τεχνικές λεπτομέρειες ε, και πολλές προτάσεις της είναι ενδιαφέρουσες. Μα και ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, θα ήθελα να σταθώ σε δύο μόνο σημεία. Σε ό,τι αφορά τη νέα αρχιτεκτονική της οικολογικοποίησης. Όντως δεν είναι αρκετά φιλοδόξη η πρόταση και θα πρέπει να συνδυάσουμε τους διάφορους μηχανισμούς για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και το οικολογικό πρόγραμμα μεριμνώντας ώστε να μην περάσουμε στο greenwashing, δηλαδή ε, να μην πέσουμε στην παγίδα της, ε, οικολογικής της οικολογικοποίησης που είχαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια. Δεν συμφωνώ με το ανώτατο όριο των 100.000. Είναι υπερβολικά υψηλό αυτό. Και πιστεύω ότι ε, καλύτερα να έχουμε ευρωπαϊκή θέσπιση κατά ανωτά των όριων και όχι εθνική γιατί θα δημιουργηθούν μεγαλύτερε διαφορές. Επίση να συμπεράλαβουμε και το κριτήριο της απασχόλησης στην κατανομή των ενισχύσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκαρσία για την έκθεσή της. Ήταν ε, πραγματικά πολύ δύσκολη ίσως είναι η πιο δύσκολη που έχουμε διαχειριστεί στη θητεία μας, γιατί μιλούμε για ε, ελλείψεις που υπάρχουν στη βασική πρόταση, ε, μιλούμε για ευελιξία, πολλά πρέπει να προσθεθούν και τώρα πρέπει να δούμε και τα στατηγικά σχέδια τα οποία πρέπει να εκπονήσουν τα κράτη-μέλη, για το αναπτυξιακό όραμα του κάθε κράτους μέλους, κυρίως για την Ήπεθρο, όπου ο, θα συνδυαστούν ο πρώτος και δεύτερος πυλώνας. Σημαντικός θα είναι ο διάλογος στα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμής ήταν και αυτός ελλειπής και λίγοι τελικά έχουν καταλάβει τι ακριβώς κάνει η γεωργία, γιατί είναι απαραίτητε κάποιε δραστηριότητε τη γεωργία και για το περιβάλλον κτλ. Και σημαντικό είναι επίση να ε, έχουμε τη στήριξη των φορολογουμένων, δηλαδή των συμπολιτών μα. Εγώ υποστηρίζω την ε, ε, προσέγγιση για τι οικογενειακέ εκμεταλλεύσεις. Για το κάπινγκ θα πρέπει όντως να συζητήσουμε κάποια πράγματα ακόμα, αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση είναι καλή. σημαντική είναι η στήριξη στους νέους αγρότες. Και εδώ να προσθέσω ότι βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε εκείνους που ε, μεταβιβάζουν τις ε, ε, εκμεταλλεύσεις τους. Επίσης, σημαντικές είναι οι νέες τεχνολογίες, η μεταλαμπάδευση της γνώσης και, αυτό, και πρέπει να, γίνει, να ενισχυθεί η πρακτική αυτή. Η ψηφιοποίηση επίσης είναι πολύ σημαντική και στις τροπολογίες θα το πούμε αυτό. Υπάρχει ένα μια σκεπτική για τους γεωργούς. Έχουμε την προσέγγιση από το Ταμείο Συνοχής, από το ίντερνετ, από άλλα ταμεία. Χωρίς όλα αυτά, η ύπεθρος δεν μπορεί να επιβιώσει. Χρειαζόμαστε ε, μια ενιαία προσέγγιση για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό πρέπει να ε, αντικατοπτρίζεται στα σχέδιά μας και γι' αυτό εγώ δεν είμαι υπέρ του κατακαιρματισμού των ε, ε, κονδυλίων για την Ήπεθρο. Πρώτο σημείο, ε, καταρχάς να πω ότι όντως μιλούμε για, τις, ε, για τους γεωργούς που κατέχουν γη, για γεωργούς που δεν, έχουν, που δεν μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις που πρέπει. Μιλούμε και για, τις, ε, για τραπεζικές υποχρεώσεις, είναι σημαντικό αυτό. Το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια αυτό το θέμα. Και ε, δεύτερον, για τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα και πώς ε, μπορούμε να διαχειριστούμε τα στρατηγικά σχέδια. Μπορούμε πάντα να πούμε ότι είναι πιο σημαντικό αυτό για τον τομέα της γεωργίας. Ε, τα κράτη-μέλη τι κάνουν ωστόσο δεν μπορεί να μην έχουμε ισότητα όπλων εδώ. Θα πρέπει να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες για όλους. Ακόμα και για το greening που είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει και με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, με την πολιτική για την προστασία της φύσης, με, ε, με το εισόδημα των ε, ε, γεωργών που θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν τη γη τους. Θέλουμε ανάπτυξη της υπαίθρου. Για το life όμως είχαμε συμφωνήσει ότι ως ε, Επιτροπή Γεωργίας ότι θα ε, υπάρξουν επενδύσει. Μετά ακούσαμε τον ε, συνάδελφο Γκερμπράντι που έλεγε ότι όλα αυτά καταργούνται πια. θα πρέπει λίγο να συμφωνήσουμε κάπου. Για την απαγόρευση τώρα νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει και θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες σχετικά για τη στρατηγική, για τις ε, πατάτες, τουλάχιστον για τις κάτω είναι πολύ σημαντική. Ε, χρειαζόμαστε καλές τιμές επίσης για τους παραγωγούς. Έχουν αναφερθεί αυτά τα σχόλια και σε άλλες εκθέσεις. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Ε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. θα πρέπει να γίνει συζήτηση. Η εισηγήτρια ε, τι μπορεί να κάνει ωστόσο. Έχει, υπάρχει το σχέδιο της νομοθεσίας από την Κομισιόν. Εγώ άνοιξα τα αυτιά μου και προσπαθώ να ακούσω προσεκτικά τις ε, παρεμβάσεις. Πολλά ακούστηκαν και συμπεριλαμβάνονται στην ε, έκθεση. Είναι πολύ καλή λοιπόν η δουλειά που έκανε ε, την, η συγγήτρια και βεβαίως σίγουρα δεν θα αποκλείσει νέες προτάσεις που θα έρθουν από εμά. Πρέπει λοιπόν να τα διαχειριστούμε όλα αυτά, να τα συνδυάσουμε. Εγώ χάρηκα για τα όσα είπε, για το χειροκρότημα που πήρε ο κύριος Ντόρφμαν αλλά αυτό το χειροκρότημα θα πρέπει να οδηγήσει και σε σωστές αποφάσεις, κυρίως για το, ε, για το κάπινγκ δεν θέλω να πω κάτι, γιατί αν πούμε ότι επιτρέπουμε να μην υπάρχει ελάχιστη πληρωμή για ένα εκτάριο, τότε ξαφνικά θα έχουμε ε, μόνο, ε, θα, θα δίνουμε μόνο επιδοτήσεις στους, ε, σε μεγάλους ε, γεωργούς και όλοι οι υπόλοιποι δεν θα παίρνουν τίποτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε σωστές ειλικρινείς διατάξεις για να μπορέσουμε να έχουμε και εμπιστοσύνη. Πώς θέλουμε να κατανείμουμε τους, τα κονδύλια μεταξύ μικρών και μεγάλων γεωργών. δεν μπορούμε να, κάνουμε την, να έχουμε την αρχή του Robin Hood εδώ, να παίρνουμε από τους πλούσιους να τα δίνουμε στους φτωχού. Ε, θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις επιδοτήσεις, με τις, με τα, επιδοτήσεις, έτσι ώστε να υπάρξει μια εσωτερική συνοχή. Μετά, για τις ε, δεσμευμένες και τις, για τις ε, ε μπορούμε να μιλήσουμε πολύ. Ο κύριος Ντόρφμαν έχει δίκιο, γιατί δεν είναι πολύ δίκαιο το σύστημα. Μιλούμε και για τα προστατευόμενα ζώα, αλλά πρέπει να έχουμε σωστή διαχείριση για τα είδη αυτά ζώων. Νομίζω είμαστε αρκετά γενναιόδοροι με αυτή την ε, παράγραφο. Για το greening, ξέρετε την άποψή μου. Εγώ ήθελα να μπει πλήρω ε, στο δεύτερο πυλώνα, γι' αυτό δεν λειτουργήσε τελικώ καλά. Έχουμε τα αιτήσια μέτρα κλπ. Γι' αυτό αυτά τα οικολογικά προγράμματα θα πρέπει επιτέλου να ξεκινήσουν για να λειτουργήσουν και για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αλλά και πάλι πολλά συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μα, η οποία τώρα θα πρέπει να προσπαθήσει να ενσωματώσει τι πάνω από χίλιε προτάσει στην πρότασή τη. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ακούσαμε όλους τους ευρωβουλευτές που ήθελαν να μιλήσουν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε και λίγο χρόνο στην εισηγήτρια για να δευτερολογήσει. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα το πρωί να διακυπηρώσουμε. Θα κάνω πάντως ό,τι μπορώ. Η έκθεση για την μελλοντική συνεργασία μας αλλά και για το Συμβούλιο είναι πολύ καλή αφετηρία. Εδώ και μήνες συζητάμε για αυτό το καινούργιο delivery model. Θέλουμε τη στροφή της ΚΑΠ προς τις επιδόσεις, προς την επικουρικότητα και προς τις ε, δυνατότητες ε, ε, ίσω της ε, γραφειοκρατία, αλλά και μέτρα για τις γυναίκε Ναι. Είναι ε, μια στροφή αυτό το οποίο έγινε, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο γιατί δεν μπορούμε έτσι να πηγαίνουμε το ένα άκρο στο άλλο. Ας ε, ακολουθήσουμε τη μέση οδό, να έχουμε και την πίτα ολάκερ για το σκύλο χορτάτο. οι αλλαγές που έγιναν στην πρώτη επιτροπή να συνάδουν με αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα, αυτά τα οποία σήμερα συζητούμε έχουν σχέση με το πι Είναι το θέμα της συγκριματοδότησης είναι το θέμα της ε, ανάπτυξης της υπαίθρου. Καλά να μην τα αναλύσω αυτά. Για να δούμε τώρα για τους στόχους. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται, τι σημαίνει αυτό που λέει η συνθήκη για τους στόχους, πώς θα είναι η γεωργία στο μέλλον, άρα να κάνουμε μια καινούργια οδηγία και να πάρουμε τέλο πάντων την ρότα της επιτευχής των στόχων. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε για τους στόχους. Ό,τι λέμε θα πρέπει να συνάδει με τους δείκτες, με το delivery model. Αφού θέτουμε στόχους, να έχουμε και τρόπο να αξιολογήσουμε την πορεία μας προς αυτόν τον στόχο ή τους στόχους. Άρα, πάντα θέλουμε βελτιώσεις και έτσι θα προχωρήσουμε έχοντας αυτά που σας είπα στο μυαλό και για τις γυναίκες. Να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε αυτή την υπόθεση. Αυτά στα πλαίσια του στόχου 8. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε έναν ad hoc στόχο μόνο για τις γυναίκες. Ε, επίσης μας λέει η συγκεντρία τι θα γίνει με το να καλύψουμε όλους τους στόχους. Τα κρατημέλια θα πρέπει να αξιολογήσουν, να ζυγίσουν τι γίνεται και με τους εννέα στόχους. Εάν θεωρήσουν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα για κάποιο στόχο και τα λεφτά πιάνουν τόπο στους υπόλοιπους, ε, τελικά ας μην προγραμματιστεί παρέμβαση για τον συγκεκριμένο στόχο, αλλά θα πρέπει να κάνουν, μια αξιολόγηση με το νέο, για το νέο σύστημα και για τους εννέα συγκεκριμένους στόχους. Τώρα για τον ε, CPR, τον κανονισμό, θετική ήταν η υποδοχή. Έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος μπορεί να προσχωρήσει εκεί και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα πιάσουν τόπο τα χρήματά μας. Και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από την εισηγήτρια θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε αυτόν τον κανονισμό εφαρμοστικών διατάξεων. Επίσης, όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον, όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και άρα γι' αυτό θα πρέπει να τα λέμε συγκεκριμένα στην πρότασή μας αλλά να προσέξουμε να μην υπάρχει στο άρθρο 92 μία τέτοια ρήτρα όπως αυτή η ρήτρα backslide. Αυτό που τελικά θέλουμε είναι να εξετάσουμε σφαιρικά το σύνολο της δέσμης μέτρων. Τι θα γίνει με την ερεσιμότητα, τον πρώτο, το δεύτερο πυλώνα και τελικά αυτό θα διαπιστώσει η αξιολόγηση κατά πόσο όλα αυτά βοηθούν στο να πετύχουμε τους στόχους μας και τελικά να προτεραιώσουμε και το περιβάλλον. Γι' αυτό μας προβληματίζει λίγο αυτή η απάλληψη της ε, για το 30% την απάλληψη επίσης του δίκτυ της ε, ε, επίδοσης. Τώρα για τα πρωτεϊνούχα είναι ο στόχος κοινό. Θέλουμε να στηρίξουμε τον τομέα. Έστω Προεδρία θα ασχοληθεί αυτή την εβδομάδα και στον πρώτο πυλώνα καλύπτουμε τα πρωτοενούχα. Καλύπτονται στα μέτρα παρέμβασης που ονομάζονται άλλοι τομείς. Θα τα συζητήσουμε με εσάς. Τώρα όσον αφορά για το κάπινγκ είναι προαιρετικό μέτρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ. Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μας υποστήριξαν. Θέλουμε να υπάρχουν ίσες συνθήκες και δίκες για όλους παντού. Να λάβουν υπόψη το κόστος εργασίας, να υπάρξει καθεστώς απλουστευμένο, ούτως ώστε όπου υπάρχει ένταση εργασίας σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις οι αγρότες να μην είναι σε εμεινευτική θέση αντί των υπολείπων. Καταλαβαίνω ότι θέλει η συγγήτρια ότι αν βγάλει τα προγράμματα του περιβάλλοντος από τη μείωση του κάπινγκ αυτό θα είναι καλό για το περιβάλλον. Αλλά την άλλη μεριά υπάρχει ο στάχος να είναι πιο στοχευμένη η υποστήριξη για τον πρώτο πυλώνα. Εδώ όμως έχουμε δύο στόχους που αντιφάσκουν προς αλλήλους. Άρα στη συνέχεια της προβληματικής θα το ξαναδούμε για να έπαιξε τη υπαίθρου και εν προκειμένου η υποστήριξη της γυναίκας θα πρέπει να προγραμματιστεί να καλυφθεί από τα κρατημέλη από τα στατικά του σχέδια αυστηρή ε, πολιτική ε, γιατί έχουμε ήδη τον κανονισμό 1305 τα κράτη-μέλη. Υπολογίζοντας την στήριξη στους γεωργούς θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα σχετικά μέτρα θα είναι αρκετά ελκυστικά ούτως όταν προσχωρήσουν σε αυτά οι γεωργοί γιατί είναι προαιρετικού χαρακτήρα. Αυτό να σιγουρεύσουν τα κράτη-μέλη ότι θα υπάρχει χαρακτήρας κινήτρου σε αυτά τα μέλη. Τώρα εδώ υπάρχει ενδεχομένως πρόβλημα γιατί αυτές οι δεν είναι συμβατές με το πράσινο κουτί, το green box του ΠΟΕ. Διπλασιάζουμε την υποστήριξή μας, έτσι. Γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, πιθανή έξοδο από το green box. Άρα να είμαστε ρεαλιτές. Μάλιστα, τώρα όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο. Είπαμε ότι έχουμε το στατικό σχέδιο για τα κράτη-μέλη και να υπάρχει, είπαμε, ενιαία αρχή διαχείριση με την οποία να συνομιλούμε εμείς ως Επιτροπή. Σχεδόν ό,τι έχει στη διάθεσή του το κράτος μέλο για να κινηθεί σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό είναι όλα σε επίπεδο περιφερειακό. Να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό περιθώριο να κινηθούν στα στεγματικά τους πλαίσια. Αυτό ισχύει και για τα μέτρα ανάπτυξη της υπέδρου σε περιφερειακό επίπεδο. Όποιος θέλει να το κάνει είναι ελεύθερος. Και τώρα όσον αφορά τις διαχειριστικές αρχές, όσον αφορά την αρχή πληρωμών, όλα αυτά θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη διοικητική και στεγνωτική παράδοση κάθε χώρας. Τώρα, είναι λίγο πρόωρο να δούμε το χρονικό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα. Χρειαζόμαστε χρόνο για να δούμε πότε θα προχωρήσουμε σε αυτά τα σχέδια. Το χρειάζονται κρατημέλη, το χρειαζόμαστε και εμείς. Αυτό χρειάζεται χρονικό περιθώριο και βασιζόμαστε στο ότι θα εγκριθεί έγκυρα ε, αυτή η πολιτική και θα μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς με το στόχο μας της πρώτης πρώτου του 2021. Εάν δεν τα καταφέρουμε το χρονοδιάγραμμα, αυτό θα δούμε πώς θα το χειριστούμε ανάλογα με το τι προβλέπει ο κανονισμός. Άρα, πώς θα κινηθούμε τώρα με συγκεκριμένη ημερομηνία που θα είναι στο απότερο μέλλον. Αυτό θα είναι λάθος μήνυμα προς τον τομέα, προς τον κλάδο. Το θέμα είναι όλοι αυτά τα μέτρα της μεταρρύθμισης να υλοποιηθούν και να φτάσουν στους αποδέκτες τους όσο γίνεται πιο νωρίς. Σας ευχαριστώ και τώρα ο λόγος στην εισηγήτρια, αλλά το πολύ 10 λεπτά παρακαλώ. Καλώς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Φυσικά τους και ηγητές, αλλά και τους λοιπούς συναδέλφους της Επιτροπής, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις τους και τα σχόλιά τους. Όλα αυτά εμπλουτίζουν την έκθεση. Και σας διαβεβαιώ πως περιμένω και τις τροπολογίες σας. Τα σχόλιά σας θα ήθελα να τα δω και με τη μορφή τροπολογιών. Η είναι ότι όλοι οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσαρμόζονται στους καιρούς, γιατί οι καιροί αλλάζουν. Και ζούμε σε μια κοινωνία όπου με την επικοινωνιακή επανάσταση δεν διαβάζουμε πια εφημερίδες, αλλά βλέπουμε τις εξελίξεις να γίνονται ραγδαία, να αλλάζουν κάθε λεπτό. Και η κοινωνία θα πρέπει να προσαρμόζεται. Μερικές φορές έχουμε και παραπληροφόρηση. Και αν ε, δεν επαγρυπνούμε και δεν ελέγχουμε τις πηγές πληροφόρησης, μπορούμε να γίνουμε θύματα παραπληροφόρησης. Είναι σημαντικό λοιπόν να προσαρμοζόμαστε στους σύγχρονους καιρούς και στις αλλαγές. Γιατί οι πολίτες παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον ε, τις αποφάσεις μα για το κοινοτικό προπολογισμό. Και μέσα στο κοινοτικό προπολογισμό, η κοινή γεωρική πολιτική έχει σημαντικό μερίδιο. Και μιλούμε για θέματα που ε, επηρεάζουν όλη την κοινωνία, γιατί μιλούμε για ασφαλή υγιεινά τρόφιμα σε προσιτέ τιμές και αυτό είναι το ζητούμενο για τους καταναλωτές. Θα πρέπει λοιπόν να επικαιροποιούμε συνέχεια τις προτάσεις μας ε, και να τις ε, παρουσιάζουμε σωστά. Και αυτή η αλλαγή του τρόπου σκέψη είναι μια ευκαιρία που μπορούμε να δράξουμε. Και μπορεί να μην γίνεται η ευκαιρία αυτή και η πρόταση όπως μας την έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάθε λεπτομέρεια, αλλά να αξιοποιήσουμε τα κοινά σημεία για να αποφύγουμε το μεγάλο κίνδυνο της επανεθνικοποίησης που τον απευχόμαστε όλοι. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συστήσουμε μία δέσμη κοινών σημείων για όλα τα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών, ώστε να μοιάζουν μεταξύ τους ό,τι αφορά μια κοινή βάση. Η κοινή βάση θα πρέπει να είναι ίδια για όλα τα στρατηγικά σχέδια. Και σίγουρα τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Φιλανδίας δεν έχουν καμία σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ανταλουσίας, για παράδειγμα, της Νοτιού Ισπανίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στους γεωπονικούς, ε, στις γεωπονικές συνθήκες, ε, τις μετεωρολογικές, τις καιρικέ, αλλά λέμε όχι στην επανεθνικοποίηση και για να την αποφύγουμε την επανεθνικοποίηση θα πρέπει να ενισχύσουμε τα κοινά σημεία των στρατηγικών σχεδίων. Αυτές είναι οι δικές μου προτάσεις. Ελπίζω εσείς με τις τροπολογίες σας να βελτιώσετε αυτά τα κοινά σημεία, ώστε να καταστήσουμε την ε, ΚΑΠ ακόμη πιο κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί θα πρέπει ε, τα στρατηγικά σχέδια να προσαρμόσουν την ΚΑΠ στους σύγχρονους καιρούς και ταυτόχρονα να αποτρέψουμε την επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, αλλά να την κρατήσουμε κοινή, κοινή γεωργική πολιτική. Και μετά από συναντήσεις που είχαμε γεωργικά συνδικάτα, διαπιστώνω ότι αυτό περιμένουν από εμά οι παραγωγοί. Γιατί αυτό που δεν θέλουν οι παραγωγοί είναι αβεβαιότητες. Δεν θέλουν καθυστερήσεις στην ΚΑΠ. Θέλουν βεβαιότητε, θέλουν μια ασφάλεια. Και αυτό μου, μου το είπαν όχι μόνο τα ισπανικά συνδικάτα, αλλά και εκπρόσωποι γεωργών και άλλων χωρών. Και έχουν τα μάτια τους οι παραγωγοί στραμμένα πάνω μας. Περιμένουν από μας ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφύλαξη του κοινού χαρακτήρα της κοινή γεωρικής πολιτικής. Και πραγματικά έχουμε τον μπαλάκι στο δικό μας γήπεδο και μάλιστα λίγους μήνες πριν τις ευρωεκλογέ. Γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε τη δέουσα ευθύνη στις αποφάσεις που θα λάβουμε για τη νέα ΚΑΠ. Άκουσα τα σχόλια, περιμένω και τις τροπολογίες. Ε, δεν μπορώ να επεκταθώ σε όλα γιατί με περιόρισε ο κ. Σεκές. Και τώρα για το κάπινγκ, τα ανώτατα όρια. Το σχολιάσατε πολύ. Το κάπινγκ είναι το μόνο θέμα για το οποίο ήμουν ε, πραγματικά ελαστική. Από όλη την πρόταση μόνο στο κάπινγκ ήμουν ελαστική. Και αυτό γιατί μετά από συζητήσει που είχαμε τον κλάδο, με τα κράτη-μέλη και με πολλού συναδέλφου, έκρινα ότι το κάπινγκ, τα ανώτατα όρια θα πρέπει να προσαρμόζονται στι διάφορε παραγωγικέ δομέ και δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα το κάπινγκ στην Εστονία και την Πορτογαλία. Στην Εστονία, για παράδειγμα, μίλησα με τον ε, Εστονό Υπουργό Γεωργίας και μου εξήγησε ότι η πρόταση του κάπινγκ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επηρέασε το 60% της επιδοτούμενης επικράτειας. Ουσιαστικά όλους θα τους επηρέαζε, 60%. Οπότε ήταν ε, δυσανάλογο το μέτρο του κάπινγκ για την Εστονία γιατί θα ισοδυναμούσε με γενικευμένο κάπινγκ για όλο τον κόσμο. Οπότε είναι λογικό να προσαρμόζεται η ΚΑΠ στις ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό και προτείνω τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε τα, τα ανώτατα όρια στις, πραγμα, στις τοπικές πραγματικότητες. Τώρα, αν το κρίνετε ε, απαράδεκτο και αν θεωρείτε ότι δεν προσαρμόζεται η πρότασή μου στους στόχους μας, τροποποιήστε την. Πάντως, το κάπινγκ, τα ανώτατα όρια, δεν είναι τεχνικό μέτρο, είναι δημοσιονομικό μέτρο. Οπότε δεν είναι στόχο των γεωργών και κτηνοτρόφων το κάπινγκ. Το κάπινγκ είναι περισσότερο στόχο των κρατών μελών, όχι των παραγωγών. Το κάπινγκ είναι ένα δημοσιονομικό μέτρο. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έχει νόημα η ελαστικότητα, γιατί δεν είναι ένα μέτρο που θα πρέπει να είναι άκαμπτο, δεν είναι ένα τεχνικό μέτρο κοινό. Αλλά είστε ελεύθεροι, αν θέλετε να τροποποιήσουμε ε, το κάπινγκ και να είναι ευρωπαϊκό, Καλώ. Πάντως, μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για δημοσιονομικό μέτρο και δεν είναι μέτρο ενίσχυσης, γιατί η, η αναδιανεμητική ενίσχυση είναι μηχανισμό βοήθειας. Στην αναδιανεμητική πληρωμή διορθώνονται κάποιες ανισότητες μεταξύ των κρατών μέλων. Προσοχή λοιπόν αν τροποποιήσετε την πρότασή μου για τα ανώτατα όρια. Και φυσικά θα πρέπει να τηρήσουμε τους γενικούς μας στόχους. Πρότεινα 20% της βασικής άμεσης ενίσχυσης να είναι αναδιανεμητική. Και θα πρέπει να γίνει μια επανισορρόπηση χάρη σε αυτή την αναδιανεμητική ενίσχυση. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει μια ανάλυση. Δεν ξέρουμε πώς η αναδιανεμητική πληρωμή θα επηρεάσει τους Γιώργους, γιατί ακόμη προϋπολογισμό δεν έχουμε. Αυτό είναι το πιο βασικό σημείο. Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι θέλουμε να πλήξουμε την απασχόληση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι αν εφαρμόσουμε ένα κάπινγκ χωρίς να λάβουμε υπόψη την απασχόληση που στις θέσεις εργασίας κάποια ε, γεωργική εκμετάλλευση δεν είναι το ίδιο με το να πλήττουμε την ίδια τη γεωργία. Και πιστεύω ότι σίγουρα τη γεωργική απασχόληση θα πρέπει να την προστατεύσουμε, όχι να την πλήξουμε. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την ποσοτικοποίηση των στόχων. Μερικοί ζήτησαν ποσοτικοποίηση των στόχων. Θέλετε να φημώσετε, να πνίξετε, να καταπνίξετε την ΚΑΠ. Θέλετε να της βάλετε φήμωτρο και να μην μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους της. Γιατί αυτή θα ήταν η άμεση συνέπεια των ποσοτικοποιημένων στόχων. Το να καταπνίξουμε την ΚΑΠ. Σε ό,τι αφορά τις περικοπές. Περικοπές στην αγροτική ανάπτυξη. Δεν ισχύουν αυτά που άκουσα δεν δέχομαι καμία δημοσιονομική περικοπή σε κανένα τμήμα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτό που ζήτησα είναι να διατηρηθεί ο γεωργικός προϋπολογισμός στο ύψος του. Δεν είμαι υπέρ καμίας περικοπής, ούτε στον πρώτο, ούτε στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Αυτό που ζήτησα είναι η διατήρηση του προϋπολογισμού, όπως και η πλειοψηφία των Ευρωπαίων Βουλευτών. Μιλήσατε για τους νέους γεωργούς. Συμφωνώ όποιο μέτρο προσελκύει περισσότερους γεωργούς στη Γεωργία είναι ευπρόσδεκτο. Και περιμένω με αδειμονία τις τροπολογίες σας. Περιμένω πώς και πώς να τις διαβάσω. Και σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, γιατί κάποιος με κατηγόρησε για το εισόδημα για τη βιωσιμότητα. Αυτό είναι ενισχυμένη ερεσιμότητα. δηλαδή σημαίνει ότι όλη η οικολογικοποίηση είναι πια υποχρεωτικό, όχι για την λήψη του 30% της βοήθειας, αλλά για να ε, λυθεί το 100%. Δηλαδή, οι προϋποθέσεις ε, του οικολογικοποίησης δεν ε, σχετίζονται με το 30% της ενίσχυσης, αλλά με το 100% της ενίσχυσης. Έτσι θα ενισχυθεί η οικολογική συνιστόσα και θα δοθεί μεγαλύτερο, μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις της ΚΑΠ. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η αύξηση των περιβαλλοντικών μας φιλοδοξιών. Και γι' αυτό το 70% των κονδυλίων ε, σχετίζεται με αυτή την βοήθεια. Και μάλιστα τώρα, τώρα μιλούμε για εισόδημα για τη βιωσιμότητα. Άλλαξε το όνομα και δεν είναι ανώδυνη αυτή η αλλαγή του όρου. Μιλούμε για εισόδημα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αλλά το 30% είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να ζητάμε 70% για να μην ε, οδηγήσουμε σε ασφυξία τους Γιώργους. Θέλουμε διαφύλαξη του εισοδήματο για να έχουμε φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους και των Γεωργών. Και μία βοήθεια στο εισόδημα θα πρέπει να αποσυνδέεται από την περιβαλλοντική απέτηση αλλά ένα υπερβολικά υψηλό ποσοστό θα διακυβεύσει τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την ισορροπία και να το λάβουμε αυτό υπόψη. Περιμένω τις τροπολογίες σας. Θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση και όποτε κρίνεται σκόπο θα προχωρήσουμε στη συζήτηση της έκθεσης για την κοινή οργάνωση αγοράς. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκαρσία. Η αποφασιστικότητα που φάνηκε από τις ε, παρατηρήσεις ε, και τη συζήτηση. Είναι πολύ καλός ιονός για την ε, δρομολόγηση αυτού του θέματος γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε και τον κοινό χαρακτήρα της ΚΑΠ, θέλουμε και μια ελαστικότητα στην ΚΑΠ. Αυτή είναι βασική στόχη και μέρημνα των στρατηγικών σχεδίων. Επίσης το θέμα των ε, ανωτάτων ορίων θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέονται με την δομή της παραγωγής. Είναι όλα αυτά σημαντικά σημεία και προέκυψαν από τη συζήτηση. Και επίσης ανταγωνιστικό θα πρέπει να είναι το κάθε στρέμμα, το κάθε εκτάριο της γεωργικής εκμετάλλευσης. Και να δούμε και το αποτέλεσμα της παραγωγής κλίμακος και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και τέλος, εγώ δεν φοβάμαι την εθνικοποίηση της ΚΑΠ. Γιατί θα συντονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ούτως ή άλλως εξασφαλίζει ένα κεντρικό συντονιστικό ρόλο. Και θέλουμε ε, και τα Εθνικά Κοινοβούλια να ελέγχουν τα στρατηγικά σχέδια και να εξασφαλιστεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στρατηγικών σχεδίων και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να είναι και για να υπάρχει μέσο ελέγχου θα πρέπει να συμμετέχουμε σε όλη τη διαδικασία ε, της εφαρμογής και του ελέγχου και θα πρέπει ο κοινοβουλευτικό έλεγχος να γίνεται και σε εθνικό επίπεδο από τα εθνικά κοινοβούλια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και φυσικά θα πρέπει να ληφθούν ε, υπόψη τα σχόλια των Εθνικών Κοινοβουλίων για τα στρατηγικά σχέδια. Και θα πρέπει αυτό να εξασφαλιστεί. Σας ευχαριστούμε. Ε, προσπάθησα να μην περιορίσω τη συζήτηση. Ε, σε όλους, παρόλο που ε, τελικά ζήτησαν το λόγο και τον έλαβαν όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 3 Δεκεμβρίου και για τις δύο εκθέσεις που εξετάσαμε σήμερα. Και μην ξεχνάτε την επιστολή του κυρίου Ταγιάννη. Διαβάστε την παρακαλώ, σας τη δώσαμε. Ευχαριστώ. Διακόπτουμε τώρα και θα τα ξαναπούμε στις 2.30 που έχουμε και εξωτερικούς καλεσμένους. Γι' αυτό σας παρακαλώ, να είστε ακριβείς, να μην έρθουν οι καλεσμένοι και εδώ να διαέθουσα. 2.30 ραντεβού.